Okay, friends, we start. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Περνάμε στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης. Ξεκινούμε με τη συζήτηση της ε, κατάστασης στην απασχόληση και τις εργασιακές συνθήκες στον ε, Ευρωπαϊκό Κλάδο της Πολιτικής Αεροπορίας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους ε, του κλάδου αυτού Χαιρόμαστε για την παρουσία σας και ανυπομονούμε για τη συζήτηση. Μάλιστα είχαμε συναντήσεις τους τελευταίους μήνες γιατί ήταν σημαντική η προτεραιότητα και του πολιτικού προγράμματος αλλά και στην επικαιρότητα μπήκε το θέμα της πολιτικής αεροπορίας και στο πρόγραμμα εργασιών των συνδικάτων. Ακούστηκε και το ζήτημα του κοινωνικού dumping στην πολιτική αεροπορία. Το συζητήσαμε και στην Επιτροπή μας, το συζητήσαμε και στην Επιτροπή Μεταφορών και στις πολιτικές μας ομάδες και παρόλο που οι βουλευτές είναι λίγοι γιατί είμαστε πέμπτη απόγευμα και πολλές επιτροπές ψηφίζουν. Πολλοί παρακολουθούν με ζωηρό ενδιαφέρον τη συζήτηση γιατί αναμεταδίδεται και μέσω του διαδικτύου. Πολλοί συμπολίτε μας λοιπόν μας παρακολουθούν και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για σύντομες εισαγωγικές ομιλίες για την κατάσταση και τις εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Γιατί περί παγκοσμιοποίησης πρόκειται τελικά. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Εμμανουέλ Γιαχάν, την Ένωση των Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιριών και πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου του Ευρωπαϊκού Κλάδου της Πολιτικής Αεροπορίας. Κύριε Γιαχάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, δώσω κάποιες γενικές γραμμές στη συζήτηση και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Καταρχήν, ε, έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Όταν οι αεροπορικέ εταιρείες δηλώνουν τους ε, εργαζομένους τους σε μία χώρα, αλλά αυτοί απασχολούνται σε άλλη χώρα, οπότε δεν πληρώνουν τις κοινωνικές φορές που οφείλουν. Μία εταιρεία που χρησιμοποιεί ε, υπαλλήλου ε, που τους δηλώνει ως ανεξάρτητους ε, ή έχουμε έναν αργοδότη με συμβάσει περιορισμένο χρόνο και ουσιαστικά πρόκειται για υπαλλήλου που όμως δηλώνονται ως ανεξάρτητοι. Άρα υπεκφεύγει ε, ο εργοδότης της υποχρέωσης καταβολής των ε, κοινωνικών επιδομάτων και εισφορών. Στο πρώτο παράδειγμα και πάλι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε ζητήσει να σας καταθέσουμε τεκμήρια. Εμείς συγκεντρώσαμε τέτοιες αποδείξεις και ειδού το αποτέλεσμα. Έχουμε ε, καταλόγους και είναι εύκολο στο εμπορικό μητρό της Ιρλανδίας. Βλέπουμε εργαζόμενους που εργάζονται μόνο για να απασχολούμενο έχουν δηλωθεί ως ε, ε, αυτοαπασχολούμενοι. Επίσης, ε, κάποιοι που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένο είδος εταιριών, τις λεγόμενες χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες. Βέβαια δεν είναι όλες, δεν βράζουν όλες το ίδιο καζάνι, μερικές τηρούν τους όρους, τους σέβονται. Αλλά οι ανεξάρτητοι κυρίως σε τέτοιου είδους εταιρείες χαμηλού κόστους εμφανίζονται. Δεύτερο παράδειγμα, χρήση σημειών ευκαιρίας και μιλούμε για πραγματικές θέσεις απασχόλησης. Έχουμε μια εταιρεία που δηλώνει τους πιλότους της, στο, στην Μπαγκόκ, ενώ ε, ε, κάνουν ε, υπερατλαντικές πτήσεις από το Gatwick με συμβάσεις ορισμένου χρόνου χρησιμοποιώντας μερικές φορές και εταιρείε αναζήτηση εργασίας, μερικές απασχόλησης με έδρα την Ευρώπη. Έχουμε εδώ αθέμητο ανταγωνισμό. Τρίτο παράδειγμα, επίκαιρο. Οι εταιρείε που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις. Μερικές μάλιστα είναι και αμερικανικές 42 δισεκατομμύρια δολάρια κρατικών ενισχύσεων έχουν λάβει. Και φυσικά αυτό επηρεάζει τη δική μας ένωση, γιατί η ΕΣΕ με την Βουλγκα Αλιτάλια, Ερμπέρλινγκ, Έτιατ και Air και με πλειοψηφικό μέτοχο την Κατάρ Airways, ως διαμαγείες, όλες τις στοιχείες μάλλον αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την ένωσή μας. Και αυτό είναι συμβολικό και ενδεικτικό της σημασίας που έχουν οι νέοι αυτοί μέτοχοι στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές. Απασχόληση, τελευταία διαφάνεια. Από το 1998 μέχρι το 2010 με βάση μια μελέτη της ε, DG Move, οι άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας ε, μειώθηκαν παρά την εμφάνιση των λόγων cost εταιριών, δεν είχαμε ουσιαστικά δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια υπάρχουν διεκιμάσεις ανάμεσα στις πόλεις και είχαμε, ενώ είχαμε αύξηση των δρομολογίων πάνω από 5% το χρόνο, ουσιαστικά δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις απασχόλησης. Τώρα έχουμε σήμερα έναν ορισμό και γνωρίζω ότι η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων είχε βοηθήσει με την θετική ε, οδηγία. Έχουμε τώρα έναν ορισμό του εργαζόμενου, της εργασίας, ε, του εργοδότη και της αμοιβή. Ορισμός υπάρχει. Εμείς οι εργοδότες θέλουμε να εφαρμόζεται κιόλας για να αποφύγουμε αυτούς τους ψευθανεξάρτητους ε, και θα πρέπει οπωσδήποτε και κατά προτεραιότητα να τροποποιηθούν κάποιοι κανονισμοί. Καταρχήν αυτοί που διέπουν ε, τις ε, κρατικές ενισχύσεις σε εταιρείε τρίτων χωρών. Επίσης, ε, αυτούς που διέπουν, τους κανονισμούς που διέπουν το Air Operator Certificate, το πιστοποιητικό των αεροπορικών εταιριών και επίσης να βελτιωθεί ο ορισμός του home base, γιατί μιλούμε για μετακινούμενους εργαζομένους Οπότε πολλές φορές ε, γίνεται κατάχρηση αυτού του ορισμού του home base. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε να τροποποιηθούν αυτοί οι κανονισμοί γιατί θέλουμε όχι λόγια του αέρα και περικοκλάδες αλλά απλά και χειροπιαστά πράγματα. Επίση έχουμε σήμερα το ναυτιλιακό τομέα. Ο ναυτιλιακό τομέα λαμβάνει κρατικές ενισχύσει. ενώ ο δικός μας κλάδος, οι αερομεταφορέ και η πλειοψηφία των αεροπορικών εταιριών έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τη φορολογία, κυρίω στις τρίτες χώρες. Γιατί εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε πολύ πιο σημαντικές επιβαρύσεις από ό,τι οι τρίτες για τις αεροπορικές εταιρείες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ελιζαμπέτα Τσίκα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών και ε, των εργαζομένων, η Επιτροπή του Θαράμου του Είμαι η Ελιζαμπέτα Κίκα Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής του Πληρώματος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών. 19.000 μέλη πληρωμάτων εκπροσωπούμε στην Ευρώπη και σκοπός της παρουσιάσεως είναι να δείξω ποιες είναι οι δυναμίες στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσον αφορά την απασχόληση στην πολιτική αεροπορία και κυρίως για τις θέσεις ε, στα αεροσκάφη του πληρώματος. Μία ενιαία αγορά δεν μπορεί να αναπτυχθεί εντός κοινωνικού πλαισίου η, η απελευθέρωση των αερομεταφορών ήταν υποφελής για τους ταξιδιώτες. Είχαν, ε, έχουν πιο φθηνά εισιτήρια να πληρώσουν, μεγαλύτερη πρόσβαση στις αερομεταφορές και αυτό το άνοιγμα στην αγορά ε, δείχνει πλήτη και τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα εργαζομένων. Λόγω της φύσης εργασίας κινείται πολύ το προσωπικό το πλήρωμα και κυβερνήτης-κυβερνήτης ε, και πλήττονται ιδιαίτερα το φαινόμενο όμως οι συνέπειες αφορούν και άλλες ομάδες του τομέα όπως και το προσωπικό εδάφους. Ε, σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε έναν κατάλογο αδυναμιών στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις προτάσεις μας. Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, οι εργαζόμενοι κατά κανόνα διέπονται από την νομοθεσία της χώρας ε, όπου εκεί θεωρούνται εργαζόμενοι. Και εκεί που έχω την έδρα το πλήρωμα, η κοινωνική ασφάλιση δεν, δεν λαμβάνει υπόψη τις έδρας της βάσης όπως γίνεται όσον αφορά τις ασφάλειες ε, το, και τις υποχρεώσεις στην πτήση. Τώρα για υπεργολαβία και ε, προσωρινή απασχόληση χρησιμοποιούν υπεργολαβία ε, σε υπερβολικό βαθμό και προσωπική απασχόληση για μεγαλύτερη ευελιξία και επίσης και μη τυπικές μορφές εργασίας γιατί δεν θέλουν να δώσουν υπεργολαβίες εκτός Ευρώπης και θέλουν να υπερκεράσουν την νομοθεσία την εργατική και να αποφεληθούν από τις διεθνείς συνθήκες εργασία. Η ΕΤΕΦ ανησυχεί διότι στο μέλλον τελικά το πλήρωμα ίσως αντικατασταθεί από εργαζομένους από μη ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, να αφορά την οδηγία την έννοια άδεια, η νομοθεσία περί μεταναστεύσεως της Ευρώπης επιτρέπει στις εταιρείες να παρέχουν λιγότερη προστασία όσον αφορά τους εργαζόμενους σε αερομεταφορές από ό,τι άλλους εργαζομένους. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζομένους από χώρες που δεν έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διαφόρους λόγους όπως για ε, γκουβερνάντες, ε, υπεύθυνου για διασκέδαση κλπ. χωρίς να εξετάζουν το ιστορικό και θέματα ασφαλείας. Ε, Λοιπόν, θέλουν να έχουν λιγότερες δαπάνες εταιρείε και λιγότερο ειδικευμένο προσωπικό στις ε, πτήσεις μακράς διαρκείας για να έχουν ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο με άλλες εταιρείε που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτοί οι εργαζόμενοι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να διέπονται από τις ίδιες συνθήκες όπως οι συνάδελφοι των κρατών μελών. Κάτι που προβλέπεται από τους νόμους που ε, ε, θεωρούν ότι ισχύει ο νόμος της χώρας της έδρας του πληρώματο. Οπότε οι μη ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκά πληρώματα δεν χρησιμοποιούνται σαν εργαλείο για να επιβάλλουν τελικά κοινωνικό ντάμπινγκ. Η οδηγία για, τον, για το εργασία δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 2000 και υπάρχει μια ανάγκη για καλύτερη πρόβλεψη, καλύτερες διατάξεις και καλύτερη προστασία του κινητού προσωπικού ε, σύμφωνα με το ωράριο εργασίας και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας και συμφιλίωσης εργασίας και οικογενικής ζωής. Όσον αφορά τις μη τυπικές μορφές εργασίας, Έχουμε χαμηλότερες αμοιβέ και συνεισφορές για την κοινωνική ασφάλιση και μικρότερη κατάρτιση που έχει συνέπειε στην ασφάλεια. Μερική απασχόληση και προσωπική, προσωρινή απασχόληση αυξάνεται το 2000 και αυτό θα οδηγήσει ότι τα πληρώματα στο μέλλον δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομούν αρκετά ούτως ώστε να καλύψουν τι χαμηλέ συντάξει. Υπάρχει πραγματική ανάκτηση, η κοινωνική προστασία να επεκταθεί και κυρίω η κοινωνική ασφάλιση και στο προσωπικό το προσωρινό του πληρώματο και να προσαρμοστεί διόντω η νομοθεσία ούτως ώστε να καλύπτονται οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως ε, προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Νομολογία. Το κοινωνικό διάλογο, η ETF, ενθαρρύνει τους εργοδότες να εισέλθω σε συζητήσει όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα για το προσωπικό και έτσι να υπάρχουν ισότιμε συνθήκε για όλου. Και τέλο, κάτι εξίσου σημαντικό, η ETF φρονεί ότι υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για τι συνθήκε εργασία όσον αφορά τι αερομεταφορέ και προτείνουμε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τι εργασίε και συνθήκε εργασία στην πολιτική αεροπορία. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τζον Χόρν, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης των Εργαζομένων στο Πιλοτήριο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. και καλημέρα σας. Καλησπέρα σας λοιπόν κυρία Πρόεδρε και αξιότιμη Ευρωβουλευτά, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε ε, να μιλήσω εδώ. Είμαι Τζον Χόρν, αντιπρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζομένων στο πιλωτήριο των ε, επαγγελματιών πιλότων και εγώ είμαι πιλότος αεροπορικής εταιρείας. Θα σα παρουσιάσω τα πορίσματα μιας πρόσφατης μελέτης για την ατυπική αυτή εργασία και τη συνέχεια που δόθηκε. Μερικά πορίσματα είναι πολύ σημαντικά και εξηγούν πραγματικά γιατί η μη τυπική αυτή μορφή απασχόληση έχει γίνει ε, ε, κανόνας σε πολλούς κλάδους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είναι ιδιαίτερα επισφαλής και επιζήμια για την αεροπορική εταιρεία. Είχαμε προβλήματα τελευταία χρόνια, αλλά προσπαθούσαν να, να μας πείσουν ότι ήταν περιθωριακό αυτό το φαινόμενο και υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία. Με την έκθεση όμως αυτή του Πανεπιστημίου της, Γα... Γάνδης φαίνεται ότι η κατάσταση έχει αλλάξει. Δεν είναι πια η εξαίρεση αλλά ο κανόνας, οπότε ήρθε η ώρα για να αναλάβουμε δράση. Ερχόμαστε λοιπόν στο κυρίως θέμα, στο ψαχνό. Μπορούμε να επισκεφτούμε τα πορίσματα της μελέτης. Ναι, γιατί ε, έχουμε ελέγξει τις απαντήσεις 10% ε, των ε, ενεργών πιλότων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε από στατιστική άποψη είναι πολύ ρωμαλαία η μελέτη και, κατα... και καλύπτει την, την πολιτική αεροπορία. Και μάλιστα οι απαντήσεις των πιλότων δίνουν πολύ σημαντικά στοιχεία και μας επιτρέπουν να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση. Βλέπω ότι ένα έξι πιλότους απασχολούνται με μη τυπικές ε, μορφές εργασίας, δηλαδή όχι άμεσα και όχι συμβατικά. Περίπου 10.000 πιλότοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται με, το, με τη μορφή αυτή. Δηλαδή χίλια ε, αεροπλάνα που πετάνε στον ουρανό ανα πάσα στιγμή ε, είναι στερεχωμένα με τέτοιο προσωπικό. Ένα στους έξι ε, ουσιαστικά λέμε, αλλά είναι πολύ πιο συγκεντρωμένα τα πράγματα. 40% των νέων πιλότων, ηλικίες 20 με 30 ετών, δεν απασχολούνται άμεσα. Και μισές ε, από τις low cost εταιρείε ε, και τους πιλότους δεν απασχολούν άμεσα τους πιλότους τους. Και 4 στους 5 πιλότους που υποτίθεται είναι αυτοαπασχολούμενοι, ουσιαστικά απασχολούνται με τέτοιες κάλπικες συμβάσεις από low cost εταιρείες. Και ε, εδώ που φαίνεται το πιο κόλθες αποτέλεσμα της ε, κατάστασης, μισή από τους αυτοαπασχολούμενους εντός εισαγωγικών πιλότους ε, λένε ότι, είναι, ότι δεν μπορούν να λάβουν υγιείς επαγγελματικέ αποφάσεις και κρίσεις, να κάνουν κρίσεις. Τώρα, τι γίνεται με τον έλεγχο πριν την πτήση. Εδώ προσπαθώ να ελέγξω όλες, όλους τους χώρους στους οποίους έχω πρόσβαση, αναζητώντα οποιαδήποτε ελάττωμα ή διαρροέ. Αν βρεθεί κάτι, ε, καλούμε ένα μηχανικό να το διορθώσει, μπορούμε να αλλάξουμε αεροπλάνο ή να χρειαστεί να κυρωθεί η πτήση. Η απόφαση όμως δεν είναι πάντα σαφής ή εμφανής. Και σίγουρα δεν είναι αυτή η έκβαση εμπορική που περιμένει ε, η εμφανη και σιγουρα δεν ειναι εταιρεία ή οι επιβάτες. Οπότε τελικά η μοναδική, βέβαια εγώ ως πιλότος είμαι αρμόδιος και υπεύθυνος για τη μοναδική αντικειμενικά απόφαση. Τώρα, σκεφτείτε αντίστοιχη περίπτωση άλλου επαγγελματία, δικαστή για παράδειγμα. Αν κανείς πήγαινε στο δικαστήριο για φορολογικό σφάλμα ή για τροχαίο ατύχημα, θα ήσασταν ικανοποιημένο ήταν ασφαλμένη ε, η απόφαση, αν δεν ήταν σωστή ακροματική διαδικασία. Τι γίνεται ένα χειρουργός που αποφασίζει να χειρουργήσει άσχετα αν πληρούνται προδιαγραφέ προδιαγραφές ασφάλειας ή ένα βουλευτή που θα πληρώνεται μόνο αν ψηφίζει ανάλογα με την κομματική πειθαρχία και κατεύθυνση. Σκεφτείτε τώρα η επιθεώρηση του αεροπλάνου να γίνεται από κάποιον που απασχολείται με συμβόλαιο μηδενικών ωρών και που πληρώνεται μόνο αν πραγματοποιηθεί η πτήση. Τι να πει αυτό ο άνθρωπο. Ναι. Ε, και πολλοί τέτοιοι πιλότε έχουν έχουν λάβει πολλά χρήματα για μόνο το δικαίωμα να κάνουν την πτήση. Μόνο έτσι ξεκινάνε. Οπότε έχουμε πολύ αμφιλεγόμενα ενάψματα που ισχύουν για πληρώματα που πρέπει να δηλώσουν ή ότι είναι άρρωστα είτε δεν είναι κατάλληλα να πληρώσουν ή ότι πρέπει να γίνουν κάποιες εξάσεις ασφάλειας. Παρόλο που ε, συχνά υπάρχει αυτή η εξάρτηση με την ε, αεροπορική εταιρεία, ιδιαίτερα όταν ισχύουν αυτές οι μη τυπικές ε, μορφές απασχόλησης. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα που δείχνουν γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η μορφή απασχόλησης στην πολιτική αεροπορία και πραγματικά είναι τελείως παράλογο άνθρωποι που έχουν τόσο υπεύθυνε για την ασφάλεια εργασίας να απασχολούνται με τέτοιου είδους γελίες συμβάσεις. Επίσης, ε, έχουμε ένα τετάρτο ένα, ε, σημαντικούς πιλότους από τρίτες χώρες που με ένα τέταρτο της τιμής απασχολούνται στην Ευρώπη. Τι γίνεται. Θεωρείτε ότι τέτοιου είδους απομόνωση αποτελεί με της ε, κουλτούρας ασφάλειας. Επίσης, είναι, υπάρχουν στοιχεία ότι η, μετά την εισαγωγή τέτοιων συμβάσεων υπάρχουν πολύ λιγότερες α, ασφάλειας και η απομόνωση τέτοιου είδους ατυπικής μορφής εργασίας ουσιαστικά δίνουν ενάψματα για φοροαποφυγή στην εταιρεία. Κάτι που θέτει σε μειονεκτική θέση από ανταγωνιστική άποψη σε άλλες αεροπορικές εταιρείες που πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Τώρα, είναι σαφή αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί τυπική μορφή απασχόληση στην εργασία, κοινωνικά, οικονομικά και θέματα ανταγωνισμού, θεμητού ανταγωνισμού. Πώ μπορούμε να τα λύσουμε, Υπάρχουν τέσσερι έννοιε και λύσει που θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Καταρχήν, να καταργήσουμε τέτοιε συμβάσει μηδενικών ωρών και πληρωμή μόνο όταν ε, πετάξει ο πιλότος Θέλουμε ένα ασφαλές επάγγελμα και γι' αυτό χρειάστηκε ένα, ένα είδος μαθητείας, μια μορφή μαθητείας. Να ενισχύσουμε την αρχή του home base που χρησιμοποιείται στην νομοθεσία. Και μάλιστα μετά την μελέτη αυτή του Πανεπιστήμιου της έγινε μια διάσκεψη για τον αριθμό των ελέγχων που γίνεται ε, και η απάντηση ήταν δεν γίνεται κανένα, ε, κανένας απολύτως έλεγχος και ουσιαστικά δημιουργείται ένα παραπέτασμα καπνού από τις αεροπορικές εταιρείε, ε, που μερικές φορές είναι οικειοθελής η υποχρέωση, οικειοθελής η δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχων. Οπότε θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοια παραθυράκια που εκμεταλλεύονται ορισμένοι. Επίσης να αποτρέψουμε τέτοια κάλπικα συμβόλαια και να βάλουμε ένα όριο για την έμεση απασχόληση, όπως έγινε και σε άλλους τομείς. Και Επίσης να έχουμε ένα τεκμήριο άμεσης ε, απασχόλησης εκτός ε, και αν αποδεικνύεται το αντίθετο με συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης να μπλοκάρουμε τις σημαίες ευκαιρίες όπου η αρχή του, του τόπου ε, πραγματοποίησης της δραστηριότητας χρησιμοποιείται που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται η, η σημαία με βάση τον τόπο της απασχόλησης και όχι για λόγους ευκαιρίας ή βολής. Και να ε, αναθεωρήσουμε τους κανόνες των θεωρήσεων για τα μέλη του πληρώματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον καθηγητή Τσάνβου Μας επισκεφτήκατε πρόσφατα και είσαστε καθηγητής ε, της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο, ε, στην επιχειρηματικό σχολείο του Κάρντιφ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Το κοινωνικό ντάμπινγκ προέρχεται από το γεγονός ε, ότι έχουμε μια ενιαία αγορά για αγαθά και υπηρεσίες, αλλά 28 διαφορετικά πρότυπα στις χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βλέπετε στον χάρτη πόσο έχουν διεισδύσει οι αερογραμμές χαμηλού κόστους στα διάφορα κράτη-μέλη. Στις μπλε χώρες έχουν διεισδύσει πάνω από 50%. Σε κάποιες χώρες δεσπόζουν οι ε, αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Και σε άλλες χώρες είναι χαμηλή η διείσδυσή τους, αλλά επιδιώκουν την ανάπτυξή τους. Στην Ιρλανδία λοιπόν έχουν τη μεγαλύτερη διείσδυση και είναι και η έδρα της Ryanair. Και όπως έχει πει νωρίτερα, όπως έχει πει στο παρελθόν ε, ο διευθυντής της Ryanair, η Ryanair καλύπτει ε, το σύνολο της Ευρώπης κάτι σαν κοινωνική ασθένεια. Η Ryanair βλέπουμε ότι αυξάνει το μερίδιο της αγοράς της ε, και προσπαθεί πάντα να βρει νέες διαδρομές σε όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο λοιπόν ξεκινάει νέες διαδρομές σε όλη την Ευρώπη προσπαθώντας να διασφαλίσει την ανάπτυξή της. Επίσης όμως σκοτώνει και περισσότερες ε, διαδρομές άλλων εταιριών. οι μη κερδοφόρες διαδρομές και ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο ε, τις σκοτώνει η Ryanair και μετά ξεκινάνε πάλι την επόμενη χρονιά. Εάν κοιτάξετε το, την ανάπτυξη της Ryanair βλέπετε ότι έχουμε ισχυρές διακυμάνσεις. Αριστερά βλέπετε ότι επιβραδύνεται η αύξηση χρόνο με το χρόνο και βλέπουμε και όλο και μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Το θέμα λοιπόν είναι πώς αντιμετωπίζει η αεροπορική εταιρεία την ζήτηση. Το κάνει αυτό εκμεταλλευόμενοι συστήματα απασχόλησης, ε, προσφέροντας επισφαλή και βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Μέσω ε, μιας εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο προσλαμβάνει πιλότους και μέσω διαφόρων λογιστών δημιουργούνται κάποιες μικρές εταιρείες οι οποίες παρέχουν ε, οι υπηρεσίες ε, πιλότων κατευθείαν στη Ryanair. Δεν υπάρχει νομικός όρος αυτοαπασχολούμενου στην Ιρλανδία, υπάρχει όμως ένας κώδικας δεοντολογίας που μας δίνει μια ιδέα των συνθήκων που ισχύουν για κάποιον αυτοαπασχολούμενο. Για παράδειγμα, αναμένεται ο αυτοαπασχολούμενος να είναι ιδιοκτήτης της εταιρεία του, να μπορεί να προσφέρει διάφορες ε, τιμές, να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορες ε, υπηρεσίες και να παρέχει μόνος του την ε, ασφάλεια του. Δεν υπάρχει λοιπόν νομική ορισμός. Υπάρχει μόνο ένας κώδικας πρακτικής που μας δίνει τις συνθήκες που μπορούμε να αναμένουμε να ισχύουν για κάποιον ε, αυτοαπασχολούμενο. Α πάμε στην Ισπανία λοιπόν. Έχουμε εδώ πέρα έναν νέο πιλότο. Μπορεί να είναι Ισπανό, μπορεί να είναι Λετωνό, μπορεί να είναι από οπουδήποτε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει έδρα την Ισπανία. Εργάζεται με Ιρλανδικό συμβόλαιο μέσω μια εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να πετάει σε κάποια χώρα όπου προσπαθεί η Ryanair να ε, διευρύνει τις δραστηριότητε της. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, έχει λοιπόν ένα συμβόλαιο αυτοαπασχολούμενου, όπου ο κώδικας πρακτικής να λέει ότι μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε διάφορες ε, επιχειρήσεις, ε, να μπορεί να ελέγχει την δουλειά του και να φροντίζει ο ίδιος για την ασφάλισή του. Εάν κοιτάξετε όμως τη σύμβασή του, εργάζεται άμεσα για την Ryanair, την ε, στολή και την ε, ταυτότητά του την, της παρέχει η Ryanair και η Ryanair αποφασίζει πώς και πότε θα εργαστεί ο πιλότος. Αυτό λοιπόν σαφώς είναι ένα ε, πλαστό, ένα ψευδές συμβόλαιο αυτοαπασχόλησης, διότι δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια. Το συμβόλαιο μπορεί να λέει ότι είναι συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να λέει ότι αν ο πιλότος δεν μπορεί να παράσχει την εργασία θα πρέπει να βρει αναπληρωτή. Αυτό όμως είναι το λεγόμενο συμβόλαιο boilerplate. Ένα συμβόλαιο το οποίο να μην μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στα μέρη. Αναρωτηθείτε λοιπόν το εξής. Ο πιλότος μπορεί να φέρει κάποιον αντικαταστάτη. Εάν ο πιλότος δεν μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες κάποια συγκεκριμένη μέρα, είναι άρρωστος, έχει άλλες δεσμεύσεις. Ένας αυτοαπασχολούμενος ε, θα μπορεί να βρει αντικαταστάτη. Ε, οι περισσότεροι ε, οι υπάλληλοι λαμβάνουν το πλάνο εργασίας τους τελευταία στιγμή και θα πρέπει βέβαια και το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει να συμμορφώνεται με τους κανόνες περί περιορισμού χρόνου πτήσης. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν για ένα πιλότο συνήθως να βρει αντικαταστάτη. Δεν, δεν πληρούνται λοιπόν οι προϋποθέσεις για τους αυτοαπασχολούμενους με ένα τέτοιο ε, συμβόλαιο. Τι γίνεται σε χώρες που έχουν τελείως διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. Ε, μάλλον όλοι γνωρίζουμε το δανέζικο μοντέλο του ε, flexicurity, της ελαφασφάλειας. Ξέρουμε ότι παρέχονται πολύ ψηλά κοινωνικά πρότυπα, πολύ καλές θέσεις εργασίας, βασίζεται στην ευελιξία, στις ενεργές πολιτικές αγοράς εργασίας και στην κοινωνική προστασία. Αυτά όμως παρέχονται κυρίως μέσω μιας συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Δεν παρέχονται από το δίκαιο περί απασχόλησης. Εάν λοιπόν η Ryanair θέλει στην ε, Δανία να εργαστεί εκτός συνδικάτων, που είναι η πολιτική της εταιρείας, τότε πώς θα προστατεύονται οι εργαζόμενοι, διότι ε, τα, περισσότερα από αυτά τα δικαιώματα προέρχονται από τις συλλογικές συμβάσεις ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργοδότες. Ε, το μοντέλο της Ράνια λοιπόν προκαλεί σημαντικά προβλήματα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να αναρωτηθεί λοιπόν. Επιτρέπεται το, ε, το rule shopping, το να αναζητάει κανείς ε, το, ε, τους ευνοϊκότερους κανόνες, είναι βιώσιμο το μοντέλο αυτό και είναι ασφαλές. Ακούσαμε ήδη τους πιλότους και τις ανησυχίες τους σχετικά με την ασφάλεια. Και αν θέλουμε να ρυθμίσουμε τον τομέα αυτόν, θα πρέπει να εξετάσουμε ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να συμμορφώνεται με την ανταγωνιστή οικονομία της κοινωνικής αγοράς. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κινητικότητα των κεφαλαίων στον τομέα της αεροπλοείας και θα πρέπει να εξετάσουμε πώς εφαρμόζονται τα κοινωνικά πρότυπα στις διάφορες χώρες. Διότι εάν προσλάβουμε κάποιον ως αυτοαπασχολούμενο με Ιρλανδικό συμβόλαιο και αυτό δεν συμμορφώνεται με τον εθνικό σας κώδικα, τότε σαφώς χρειάζονται καλύτεροι κανόνες ε, ε, εφαρμογής σε, σε εθνικό επίπεδο. Όλους αυτούς τους κανόνες θα πρέπει να του εξετάσουμε σε ευρωπαϊκά συμβόλαια όπου διαπιστώνεται ότι γίνεται κοινωνικό dumping και αναζήτηση των ευνοϊκότερων καθεστώτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντόρκ Γκίλη, συντονιστή διεθνούς, του Ινστιτούτου Διεθνούς Ερεύνας για τις κοινωνικές απάτες και τον Λίαν Βάλκε που είναι ειδικό το Διεθνές Αυτό Ινστιτούτο. Έχετε λοιπόν το λόγο, καλώς ήρθατε κιόλα. Θα σας οδηγήσω σύντομα μέσω στη μελέτη που έχουμε φτιάξει. Είναι στο διαδίκτυο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Πρώτα απ' όλα, κάναμε μια πιλωτική μελέτη των μορφών άτυπης εργασίας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και συλλέξαμε στοιχεία, κάτι που έλειπε, η μελέτη αποτελείται πρώτα απ' όλα από έρευνα μέσω υπολογιστή του, εκαναμε συγκριτική έρευνα στοιχείων που υπήρχαν. Κάναμε λοιπόν σύγκριση των στοιχείων που συλλέξαμε, το ανέφερε αυτό ο Τζον. Συνολικά πήραμε πάνω από 6.633 απαντήσεις από άτομα διαφορετικών υπηκότητων που αυτοί εργαζόταν σε διάφορους τομείς της πολιτικής αεροπορίας κυρίως σε, αεροπορικέ σε αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και δικτύου και διάφορες λοιπόν αεροπορικές εταιρείες, διάφορα είδη απασχόλησης. Ο Τζον είπε ήδη ότι στη μελέτη μας το βασικό, οι περισσότεροι μας είπαν μάλλον ότι είχαν άτυπες σχέσεις εργασίες ε, βλέπετε ότι 79 ήταν άμεσα, 79% ήταν άμεσα απασχολούμενοι και 16% ε, έμεσα Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα, ήδη ο Τζον είπε ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα, διότι αυτοί που εργάζονται μέσω μη τυπική απασχόλησης βρίσκονται σε συγκεκριμένους τομείς και ηλικιακέ ομάδες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί ήδη αναφέρθηκε σε αυτά τα θέματα ο Τζον. Οι νεότεροι με μικρότερες εμπειρίες έχουν περισσότερες πιθανότητες να μπουν σε αυτή τη μη τυπική απασχόληση. Μπορώ να σας δείξω τι σημαίνει κάτι τέτοιο η άτυπη απασχόληση. Ε, δηλαδή, η εταιρεία απασχολεί διάφορα μέλη του πληρώματος και όλοι έχουν βάση σε μια χώρα. Ουσιαστικά είναι η χώρα έδρα της αεροπορικής εταιρείας. Γίνεται πιο δύσκολα η κατάσταση όταν έχουμε ενδιάμεσο και ακόμα πιο δύσκολο αν χωρίζεται διάμεσος φορέας μεταξύ μιας υπηρεσίας προσωρίνη απασχόλησης και κάποιου διάμεσο λαβητή αν θέλετε ε, και μετά έχετε διάφορες άλλες συνθήκες, διάφορες καταστάσεις πιο περίπλοκη κατάσταση είναι αυτή όπου διάφορες θηγατρικές δημιουργούνται σε διάφορες χώρες, όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Τι ανακαλύψαμε λοιπόν. Υπήρχε μια, ένας διαχωρισμός αγοράς εργασίας, απομόνωση. Οι νεότεροι πιλότοι με μικρότερη εμπειρία έχουν περισσότερε πιθανότητε να μπουν σε μια μη τυπική μορφή απασχόληση. Ε, είδαμε επίσης ότι υπάρχει και κάποιο κίνητρο για τη μείωση του κόστους και προσπάθεια για τη μείωση του κόστους με προσλήψεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μέρος του πληρώματος που κοστίζει 100 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κόστιζε 65 ευρώ στην Ταϊλάνδη και 35 στην Κίνα. Και μπορείς, άμα ψάξεις, να βρεις και πιο φθηνός. Όπως προανέφερα λοιπόν, είδαμε ότι στην αρχή της καριέρας ένας πιλότος ο οποίος έχει χρεωθεί, διότι κοστίζει η εκπαίδευσή του, του κοστίζει κάτι ανάμεσα στα 80.000 και 120.000 ευρώ η εκπαίδευσή του και θα έχει λιγότερες πιθανότητες να προσληφθεί από μια ομάδα δικτυού ε, και πιο πιθανό είναι να τον προσλάβει μια εταιρεία χαμηλού κόστους. Όμως υπάρχουν κάποιοι όροι. Μη τυπικό δεν εντοπίζεται μόνο στα ψεύτικα συμβόλαια ε, ίσως αφορά και το ποσοστό της ευελιξίας, κάτι που απαιτούν βασικά εργοδότες και κυρίως οι εταιρείε χαμηλού κόστου και σε λιγότερο βαθμό ε, οι εργαζόμενοι, αλλά καμία φορά συμβαίνει και αυτό. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Κοινωνικά και φορολογικά κόλπα. Προσπαθεί να βρει το πιο βολικό νόμο η εταιρεία, να βρει την πιο φθηνή χώρα για να πληρώσει τις κοινωνικές εισφορές ε, και τους φόρους τους χαμηλότερους. Πολύ συχνά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο εργοδότης να εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία και έτσι δημιουργείται ανασφαλής ε, ε, απασχόληση και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ αεροπορικών εταιριών ταυτόχρονα. Τώρα, αυταπασχολούμενος πιλότος Μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Αμφισβητούμενο, συζητήσιμο, ποικίλουν οι απόψει. Όμως, ξανά, ένας πραγματικά αυτοπασχολούμενος πιλότος πρέπει να διαχωριστεί από εκείνον ο οποίος είναι αυτοπασχολούμενος, ψευδό αυτοπασχολούμενος. Η ψεύτικη αυτοπασχόληση είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί, διότι η αυταπασχόληση και αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα πρέπει τώρα να θυμηθούμε ότι η νόμιμη υπεργολαβία είναι κάτι που είναι διαφορετικό από τις ψεύτικες αλυσίδες υπεργολαβίας. Η πολιτική αεροπορία, μην το ξεχνάμε αυτό, έχει μορφές υπεργολαβίας, παραδείγματος χάρη μίσθωσης που είναι νόμιμη η μίσθωση, και ξεκινάει το πρόβλημα και χρησιμοποιείται σε αυτέ τι αλυσίδε υπεργολαβία τη ψευδή. Άρα έχουμε πρόβλημα μεταξύ νόμιμη υπεργολαβία και παράνομη ψεύτικη, α πούμε, εικονική. Και ποιο είναι αυτό ο εικονικό, ο ψεύτικος ε, εργοδότη. Λέμε ποιο είναι ο ψεύτικος αυτοαπασχολούμενο. αλλά αρχίζουμε και βλέπουμε καταστάσει όπου έχουμε εικονικού εργοδότε. Δηλαδή μέλη πληρώματο τρίτη χώρα προσλαμβάνονται έχοντας ελάχιστη ε, κοινωνική προστασία, μένουν εκτός της νομοθεσίας που τους προστατεύει εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως κλπ. κλπ. Ένα από τα βασικά σημεία και βασική ανησυχία είναι ότι μια άτυπη απασχόληση δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο εξάρτησης. Το προανέφερα αυτό. Και αυτή η εξάρτηση έχει αντίκτυπο. Όσον αφορά τις δυνατότητες και την προθυμία των μελών του πληρώματος ή του κυβερνήτη να, να, να λάβει αποφάσεις ανεξάρτητες όσον αφορά την ασφάλεια. Αν δείτε την έκθεση θα δείτε κάποιες ενδείξεις ε, και κάποια στοιχεία σχετικά με αυτό. Τώρα ερωτήσεις. Τι θα κάνουμε όσον αφορά την έρευνα που κάνουν οι εταιρείε για να βρουν τη πιο φθηνή, τη βολική νομοθεσία. Ε, υπάρχουν ισότιμες συνθήκες στις αερομεταφορές δεν μιλάμε μόνο για συνθήκες ευρωπαϊκές, αλλά παγκόσμιες. Ήδη αναφέρθηκαν διάφορα παραδείγματα αυτού. Μία από τις λύσεις που αναφέρθηκε ήταν να βρούμε νέες διασυνδέσεις. Κάτι που δεν είναι εύκολο. Διότι διάφοροι τομείς της νομοθεσίας και διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται αναλόγως και τονίζω μέλη του πληρώματος σε άτυπες μορφές εργασίας έχουν το κίνδυνο, δηλαδή έχουν το κίνδυνο να βάλουν προτεραιότητα όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα και στην ασφάλεια και τα θέματα της ασφαλείας ε, υπονομεύονται έτσι. Και όπως είπε και ο Τζον, έχουμε θέματα εφαρμογής νομοθεσίας, ελέγχου, χρειάζεται κατεπηγόντως να υπάρχει ε, συνεργασία διασυνοριακή, πολυτομιακή και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των ε, αρχών ελέγχου και επιθεώρησης. Κάποιες, ε, τε, κάποιοι φορεί θα πούν ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά η έκθεση δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια και τη συνεργασία. Και κάτι άλλο που δεν πρέπει να λησμονούμε είναι η νοτροπία της διοίκησης. Κάποιες νοτροπίες δεν ταιριάζουν με τα ασφαλή συστήματα διαχείρισης των αεροπορικών εταιριών και των πτήσεων γενικότερα. Ε, και ένα από τα σαφή συμπεράσματα της εκθέσεως είναι ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν είναι το δέον ε, που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες πρακτικές και στα μοντέλα τα επιχειρηματικά λύσεις. Έχουμε κάνει διάφορες συστάσεις. Ε, μία από αυτές διεύρυνση, αύξηση των κανονισμών όσον αφορά τις σχολές ε, ε, που πηγαίνουν τα πληρώματα και υποχρεωτική μαθητεία ε, και πώς μπαίνουν υποψήφοι καινούργοι, τα καινούργια μέλη του πληρώματος στην αγορά εργασία. Ποιο είναι, ποιος είναι ο μοναδικός παράγων, είναι ο κανόνας της βάσης που προσπαθεί αυτός ο κανόνας της βάσης να διορθώσει προβλήματα του παρελθόντος αλλά υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τον κανόνα της βάσης, περιγράφονται στην έκθεσή μας τα προβλήματα και θα πρέπει να εξεταστούν. Ολοκληρωμένη πολυτεμιακή ε, προσέγγιση είναι κάτι που απαιτείται και όχι μόνο αναθεωρώντας το νομικό πλαίσιο, αλλά και συνεργαζόμενοι στην εφαρμογή των μέτρων και την επιβολή του νομικού πλαισίου. Και είπαμε σαφώς ότι είναι κοινή πάλι όλων των ενδιαφερομένων αυτή. Λοιπόν, ένα από τα σχόλια που κάναμε είναι και το εξή. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι πρέπει να συνεργαστούν. Α μην περάσουμε τα ίδια που πέρασαν και οι θαλάσσιοι μεταφορές, διότι αυτό βλέπουμε σήμερα. Και πέρασα τα μεσάνυχτα ήδη, ήδη έχουμε καθυστερήσει με άλλα λόγια. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει και η κυρία Βάλκε να προσθέσει κάτι. Όχι. Ευχαριστώ. Βλέπω δύο συντονιστές. Οπότε έχετε το λόγο αν θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις ή να προσθέσετε κάτι. Κυρία Στάινρουκ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ όλους όσους μας έδωσαν σημαντικές αλλά και ανησυχητικές πληροφορίες και στοιχεία σήμερα. Βλέπουμε εδώ έναν πόλεμο τιμών στον διεθνή ανταγωνισμό και χρειαζόμαστε επιγόντως ευρωπαϊκές προϋποθέσεις πλαίσιο. Και καλό θα είναι να έχουμε και διεθνή πρότυπα όπως υπάρχουν σε άλλους τομείς. Συμφωνείτε? Και το ερώτημα για μένα είναι ότι οι καταναλωτές είναι συχνά το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες και οι σχετικές υπηρεσίες για να προωθήσουν ακριβώς τέτοιες εξελίξεις. Πιστεύετε ότι είναι σωστό επιχείρημα ότι οι καταναλωτές κοιτούν μόνο την τιμή στο εισιτήριο και δεν ασχολούνται με το ποιος βρίσκεται στο κόκπιτ. Και εάν είναι τόσο ακριβή η εκπαίδευση του πιλότου, και υπάρχει και Επιπλέον εξειδίκευση για κάποια αεροσκάφη που στοιχίζει ακόμα περισσότερο, μιλάμε για 200.000 ευρώ, πάνω από 200.000 ευρώ για την εκπαίδευση. Τότε έχει όντως και το θάρρος ο πιλότος να κάτσει σπίτι του τη στιγμή που οικονομικά εξαρτάται από μια τέτοια σύμβαση. Έχετε εμπειρίες από αυτό και από το πώς έχουν εξελιχθεί για παράδειγμα οι άδειε ασθενεία. Οι εταιρείε που πετούν εντός της Ευρώπης. Διαπιστώνεται ότι όλες συμμορφώνονται με τους κανόνες, ε, διότι νομίζω ότι υπάρχουν εταιρείε εκτός Ευρώπης, ε, μάλλον ευρωπαϊκές εταιρείε που όταν πητούν εκτός Ευρώπης ε, εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες. Μας δώσατε πολύ υλικό να εξετάσουμε στο σπίτι μας. Ο κύριος Τέρνμπουλ είπε ότι η Ryanair δημιουργεί 200 καινούριες νέες διαδρομές τον χρόνο, αλλά ε, καταργεί άλλες 120. Μπορείτε να μας πείτε τι συνέπειες έχει αυτό στην, στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας, δηλαδή στους τομείς που εξαρτώνται από την αεροπλοεία. Και επίσης το θέμα δεν είναι μόνο το προσωπικό καμπίνα, ε, ε, έχουμε και τις υπηρεσίες εδάφους όπου υπάρχουν εργαζόμενοι στους οποίους ασκείται πίεση. Και εδώ υπάρχουν ε, ψευδός αυτοαπασχολούμενοι ή άλλοι τύποι συμβάσεων. Τίθεται λοιπόν το θέμα της ευθύνης. Είναι ξεκάθαρο το θέμα της ευθύνης. Μπορείτε να μας ενημερώσετε εάν όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν συνέπειε και για τους ε, καταναλωτέ. Σας ευχαριστώ και πάλι, Μα δώσατε πολύ υλικό να εξετάσουμε. Ελπίζω και η Κομισιόν να ασχοληθεί με το υλικό αυτό. Εμείς οι Ευρωβουλευτές σίγουρα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Έχουμε υποβάλει και κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν αλλά φαντάζομαι ότι και οι άλλοι συνάδελφοι θα έχουν να σας θέσουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως η Ειρήνα θέλει το λόγο για τους... Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις πολύ ενδιαφέρουσες αλλά και κάπως ε, ανησυχητικές ε, ομιλίες σας. Εμείς οι Ευρωβουλευτές ε, χρησιμοποιούμε πολύ τα αεροπλάνα και γι' αυτό μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό όχι μόνο από θεωρητικής πλευράς ε, αλλά και από πρακτικής. Ε, γνωρίζετε ότι είμαι Δανέζα. Κάποιος ε, από τους ομιλητές αναφέρθηκε στο δανέζικο μοντέλο, αναφέρθηκε στο μοντέλο αυτό της αγοράς εργασίας. Οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις συνάπτουν τις συλλογικές συμβάσεις και από εκεί προκύπτουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και μάλιστα γίνεται αυτή τη στιγμή αγώνας κατά της, της Ryanair που θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την, τους κανόνες της αγορά αγοράς ε, της ε, Ευρώπης ε, και έτσι να αμφισβητήσει τις κινήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά της εταιρείας. Πώς μπορούμε λοιπόν να υπερασπιστούμε το σύστημα αυτό με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τη στιγμή που οι εταιρείε χρησιμοποιούν ως δικαιολογία τις άλλες χώρες όπου υπάρχει πολύ χειρότερη προστασία των εργαζομένων. Πώς μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε τους εργαζομένους μας, μια επιθυμία που έχουμε όλοι μας, ε, χωρίς υποχρεωτική νομοθεσία, διότι καταλαβαίνω ότι θέλετε νομοθεσία για να καταργηθούν οι περίεργες μορφές απασχόλησης, ε, πώς μπορούμε όμως να διασφαλίσουμε και τον αγώνα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άγνες Γιονγκέριος, ε, Αντιπρόεδρος. ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους καλεσμένους ε, για τις ομιλίες τους, γιατί μας διαφωτίζουν για δύο κυρίως θέματα. Και για το κοινωνικό dumping που πρέπει να το σταματήσουμε και το θέμα της αυτοαπασχόλησης ή των δίθεν συμβολέων ή των συμβολέων σε αυτοαπασχολούμενους. Μιλούμε για ένα κλάδο, την πολιτική αεροπορία, που και τα δύο θέματα είναι φλέγοντα. Και μάλιστα με ιδιαίτερη χαρά έμαθα ένα νέο όρο, το rule shopping, ε, την αναζήτηση της βολικής νομοθεσίας. Ε, ανακύπτει έτσι ένα νέο στοιχείο στη συζήτηση. Εγώ βλέπω δύο όψεις ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μία της όψη είναι η όψη της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, η χρηματοδότηση της μελέτης, γίνεται από αυτή για να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα των εργασιακών συνθήκων τον κλάδο σα. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η μελέτη που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπω και τη Γενική Διεύθυνση MOVE όπου όταν θέτουμε ερωτήσεις του τύπου γιατί πιστεύετε ότι αυτό που κάνει η Norwegian Air είναι αποδεκτό και αρχίζουν τα επιχειρήματα με τη σκοπιά του καταναλωτή. Γιατί μας λένε ότι οι λόγος εταιρείε εξυπηρετούν τον καταναλωτή, είναι ελκυστικές για τον καταναλωτή, αλλά θα πρέπει να προσαρμόσουν τις εργασιακές του συνθήκες. Τέτοια επιχειρήματα ακούμε. Και αυτό δεν μας βοηθάει να βρούμε λύση, γιατί έχουμε δύο διαφορετικές αντικρώμενες όψεις. Και παρακολουθώντας τη συζήτηση και ακούγοντας προσεκτικά τα σχόλιά σας και συνδυάζοντας τα με αυτό που γνωρίζω για τους ναυτικούς, για την ναυτιλία, έχουμε εκεί συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμφωνίες σε εθνικό επίπεδο ή σε εταιρικό επίπεδο. Έχουμε τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Βέβαια, εσείς δεν έχετε όπως η ναυτική βεβαια εσεις δεν εχετε από συναυτική μια ειδική ναυτιλιακή σύμβαση, αλλά ίσως θα μπορούσατε να διεκδικήσετε για να συστηθεί στη στο ΔΟΕ μια ειδική επιτροπή που θα ασχολείται με την πολιτική αεροπορία, με τις αεροπορικές εταιρείε. Και έχουμε και τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα άλλο επίπεδο, και έχουμε και την ενωσιακή νομοθεσία, τις νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διερωτώ λοιπόν, Ποιο επίπεδο κατά τη γνώμη σας υπερτέρει. Πώς θα πρέπει καταρχήν να αντιμετωπίσουμε το θέμα, πού θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Πρώτα να ενισχύσουμε τα συνδικάτα στις συλλογικές τους διαπραγματεύσεις με τις αεροπορικές εταιρείες. Ή να περιμένουμε περισσότερα από τις παρεμβάσεις της νομοθετικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν ναι, πώς αντιμετωπίσω αυτή τη σχιζοφρένεια μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων Απασχόλησης ε, Μεταφορών. Για το ίδιο θέμα έχουμε τελείως αντικρώμενες ε, συμπεριφορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από δύο διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις. Ευχαριστώ κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες. Όπως ήδη είπαν οι συνάδελφοι, ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που ακούσαμε. Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια επίκριση. Βρίσκω θλιβερή την τόσο μικρή συμμετοχή των Ευρωβουλευτών για ένα τόσο σημαντικό θέμα, μια απλή καθημερινή. Βρίσκω ότι είναι πολύ περίεργο το ότι είναι τόσο λίγοι οι ευρωβουλευτέ. εδώ. Πιστεύω ότι ο καθένας μας θα πρέπει να κάνει λίγη διαφήμιση εντός ε, της κάθε πολιτικής ομάδας. Θα μου πείτε εντάξει, είναι θέμα που αφορά όλες τις ε, πολιτικές ομάδες. Όπως και να έχει, η αεροπλοεία είναι πολύ ευαίσθητος τομέας από πλευράς ασφάλειας και αυτό μου προκαλεί ανησυχίες. Εγώ εδώ και 20 χρόνια εργάζομαι στον τομέα των οδηγικών και σιδηροδρομικών μεταφορών και συγκρίνω με τις συνθήκες που έχουμε εκεί. Σιγά σιγά προσπαθούμε να θεσπίσουμε και να εφαρμόσουμε κανόνες. Η κατάσταση βελτιώνεται αν και δεν είναι ιδανική. Εδώ όμως βλέπουμε το αντίθετο. Έχουμε έναν πολύ ευαίσθητο τομέα από πλευράς ασφαλείας με ικανοποιητική ρύθμιση, αλλά η ποιότητα των θέσεων εργασίας ε, ε, επιδεινώνεται και έτσι μειώνεται και το επίπεδο της ασφάλειας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που με ανησυχεί. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν η ρύθμιση που αφορά την έδρα. Όσον αφορά λοιπόν την έδρα των εργαζομένων, την έδρα βάσης, εγώ θα έλεγα ότι είναι περιττή. Ουσιαστικά ακυρώνεται από τις αεροπορικές εταιρείες τη στιγμή που δρούν εκτός Ευρώπης και βρίσκουν πάντα τρόπους να παρακάμπτουν αυτόν τον κανόνα. Επιπλέον, όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο, πάντα καταλαμβάνουμε προσπάθειες να βελτιώσουμε τον διάλογο. Και γνωρίζω ότι διάφορες οργανώσεις, συνδικαλιστικές και άλλες, εκπροσωπούνται στον κοινωνικό διάλογο. Εσείς πώς βλέπετε τις καθημερινές εργασίες στον κοινωνικό διάλογο. Έχετε εδώ... Ε, ε, ακούτε εδώ πολλά παράπονα χωρίς να υπάρχει πρόοδος. Επίσης, ε, όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας, δεν έχω ε, εικόνα για το θέμα αυτό. Από τη μία μειώνονται οι θέσεις εργασίας, από την άλλη ε, βλέπουμε όλο και περισσότερες στήσεις. Δηλαδή έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας. Αλλά αυτό πόσο μπορεί να συνεχιστεί, πόσο μπορεί κανείς να τεντώσει το σκηνή πρώτου να σπάσει. Είναι και αυτό κάτι το οποίο βλέπω πολύ επικριτικά. Και μια προσωπική ερώτηση. Όσον αφορά τις εθνικές αρχές ρύθμισης, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις προσφυγής των αρχών κατά αεροπορικών εταιριών. Ε, όλα αυτά περιορίζονται σε μια επίπληξη ή ε, έχουν και συνέπειες. Έχει η ΕΑΣΑ τη δυνατότητα όχι μόνο να ελέγχει αλλά και να επιβάλλει κυρώσεις. Μια προσωπική ερώτηση είναι αυτό από πλευρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ είμαι συντονίστρια στην Επιτροπή Μεταφορών και το θέμα αυτό της πολιτικής αεροπορίας ε, και του κοινωνικού ντάμπινγκ ε, μας ενδιαφέρει όχι μόνο στην πολιτική αεροπορία, είναι μάστιγα και στις οδικές και στις ε, θαλάσσιες και στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Σας ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε, για τις παρουσιάσεις σας. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη έχει και κάποια ευθυνούλα, γιατί βρισκόμαστε σε μια ξέφρενη κούρσα απελευθέρωσης των περισσότερων κλάδων αλλά η αδυναμία των κοινοτικών ε, κανονισμών και ρυθμίσεων ε, επέτρεψε τη δημιουργία τέτοιων πρακτικών κοινωνικού ντάμπινγκ. Οι αεροπορικέ εταιρείε ανέπτυξαν διάφορε στρατηγικέ που είναι σκανδαλώδε πραγματικά. Ε, για παράδειγμα, οι ψευτοαπασχολούμενοι, τα δίθεν συμβόλαια, Επίση, δίθεν αποσπασμένοι, ψευτοαποσπασμένοι και ε, ψεύτικες έντρες βάσεις. Και το θέμα των ψευτοαπασχολούμενων το διαπιστώσαμε στη ΡΑΕΝΕΑΡ, που το πάνω το, από το 70% των πιλότων της τους προσλαμβάνει μέσω κάποιων μικροεταιριών και 60% των αεροσυνοδών ε, προέρχονται από πρακτορία προσωρινής απασχόλησης. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Ιρλανδικής Ryanair. Αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν τελικά και από άλλες επιχειρήσεις. Οπότε βρισκόμαστε το φλέγον ζήτημα των κοινωνικών επιβαρύνσεων και των εργοδοτικών επιβαρύνσεων. Υπάρχουν κανόνες που ισχύουν, αλλά δεν εφαρμόζονται. Γιατί? Γιατί δεν διενεργούνται επαρκείς έλεγχοι. Πρώτη ερώτηση. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το καθεστώς του αυτοαπασχολούμενου Επίσης, ε, οι αεροπορικές εταιρείες σήμερα, ε, οι ανταγωνιστικές, ε, δεν είναι μόνο οι αμερικανικές, κυρίως οι εταιρείε του πεσικού κόλπου ασκούν ανταγωνισμό αθέμητο γιατί υποφελούνται από δικές τους κρατικές ενισχύσεις. Ήμουν αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στον χώρο εργασίας. Και σας διαβεβαιώ, συνάδελφοι, ότι το κοινωνικό dumping ε, ε, ισχύει και για τις εργασιακές συνθήκες. Γιατί ένας πιλότος ή ένα πλήρωμα που είναι ένα ε, κουρασμένο και αχωμένο, δημιουργεί κίνδυνο για τους επιβάτες. Και οι περισσότεροι πιλότες 20 30 ετών δεν έχουν πραγματικές συμβάσεις με τις αεροπορικές εταιρείες. Μερικές low cost εταιρείες ε, πληρώνουν ε, τους ε, πιλότους τους με τις ώρες πτήσης, κάτι που είναι σκανδαλώδες. Επίσης, η ΕΑΣΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας, πρότεινε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ασφάλεια να έχουμε γυναίκες αεροσυνοδούς που πετάνε μέχρι και στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης. Αυτό είναι μια πραγματική προσβολή και καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των γυναικών και ε, της υγείας τους. Κατά τη γνώμη μου, τέτοιες ε, γυναίκες έγκυες δεν μπορούν να πετάξουν κανονικά. Πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους. Οπότε τους λένε οι εταιρείε είτε θα πετάξετε και θα κάνετε τις δουλειά σας, είτε μπείτε σε αναρωτική άδεια, αν δεν θέλετε να πετάξετε όντας έγκυες. Οπότε βλέπουμε τι τεράστια πίεση ασκείται στο πλήρωμα της καμπίνας και στους κυβερνήτες. Δημιουργείται έτσι ένα κλίμα ε, αρνητικό για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Οπότε αυτό που σας ζητώ, εγκατακλείδη, είναι ε, να σας πω ότι στην Επιτροπή Μεταφορών έχουμε ένα πακέτο για τις αεροπορικές μεταφορές. Ερωτώ λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα δύο-τρία απολύτως απαραίτητα μέτρα για να μπούμε στο σωστό δρόμο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νταβρίλο. Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι λακωνικότατος. Συμφωνώ με αυτά που είπε συνάδελφος, κυρίως τα μέλη του ΕΛΚ όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές του θέματος. Θα είχα μια συγκεκριμένη ερώτηση να θέσω προς τον κύριο Μανουεζό που μίλησε πρώτος αναφέθηκε σύντομα στην Αμερικανική έκθεση για τον αθέμητο ανταγωνισμό των αεροπορικών ταιριών του κόλπου είναι πολύ σημαντικό θέμα προς διότι έχει αυτό αντίκτυπο για πιο παλιές ευρωπαϊκές εταιρείες που προσπάθησαν για να είναι ανταγωνιστικές να εφαρμόσουν κάθε δυνατόν μέσον για να ξεπεράσουν τα όρια και τα εσκαμμένα ούτω ώστε να διατηρήσουν την οικονομική του ισορροπία. Θα ήθελα λοιπόν να το αναλύσουμε περισσότερο αυτό, να μας πείτε κάποια πράγματα όσον αφορά αυτή την έκθεση και τι συνέχεια μπορούμε να δώσουμε. Να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιληφθεί του θέματος, που είναι θέμα του ανταγωνισμού και όπως έλεγε και η συνάδελφος ε, Καρέν ε, Μαντελή, έχει και αντίκτυπο στις, λόγω των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στις χώρες του κόλπου. Όταν οι συνάδελφοι κινούνται κατά των κρατικών ενισχύσεων, ε, πάντα συμφωνώ με τους συναδέλφους, διότι δεν ήθιστε αυτό να πραγματοποιείται στην Ευρώπη, να χορηγούνται οι κρατικές ενισχύσεις. Γιάννης Νίλσον, Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και είμαι μέλος και της Επιτροπής Μεταφορών. Και όπως υπόθηκε, θα συζητήσουμε ένα πακέτο για τις αεροπορικές, όπου συμπεριλαμβάνεται και η εντολή της ΕΑΣΑ. Και θα εξετάσουμε και τη σχέση ανάμεσα στην ΕΑΣΑ και τις εθνικές αρχές, διότι εδώ υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου όταν θα εξετάσουμε την εντολή της ΕΑΣΑ. Το βασικό ερώτημα είναι τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στις μορφές απασχόλησης, τις ευφυείς επιχειρηματικές λύσεις και την ασφάλεια στις πτήσεις. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό όταν θα το ξανασυζητήσουμε ε, αργότερα εντός του έτους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μαρτέν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη του πάνελ που πήραν το λόγο και εκείνους που μιλήσαν συναδέλφους. Και ήταν, είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέμε αλλά και τρόμαξα. Έμαθα ότι 10 με 30% των κυβερνητών και των πλοηγών, των αεροσκαφών και του προσωπικού εδάφους είναι θύματα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Κάτι που προέρχεται από την παγκοσμιοποίηση λοιπόν, που αγαπητοί συνάδελφοι, η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης ε, ήταν κάτι που υποστηρίζατε και εγκαθιδρύσατε τελικά και παγιώσατε. Ξέρουμε ότι ένας ευρωβουλευτής κατά μέσο όρο πρέπει να πάρει δύο φορές το αεροπλάνο την εβδομάδα κάθε ευρωβουλευτής. Και εγώ σκέφτομαι του επιβάτες ο πρόεδρος αντιπρόεδρος του Συνδικάτου των Κυβερνητών εξήγησε ότι έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο κατάσταση που κάποιοι κυβερνήτες δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία των αεροσκαφών που απογειώνονται. Είμαι επιβάτης, ανησυχώ, σχεδόν φοβάμαι. Λοιπόν, τι να πω. Θα κοιτάξω τα ωράρια του τρένου, θα το πω εν είδη Θα κοιτάω τα τρένα αλλά θα ήθελα να μας δώσετε πραγματικές λύσεις. Κάτι πρέπει να γίνει. Εκατομμύρια επιβάτες αφορά κάθε χρόνο και κάθε, κάθε μήνα και κάθε χρόνο αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μπενεφά, έχει ζητήσει το λόγο. Όχι. Καλώς λέει η Πρόεδρος. Θα επιστρέψουμε λοιπόν σε εκείνους που ελπίζω θα μπορέσουν να δώσουν μία, δύο ή τρεις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Και πιστεύουμε και διευθανόμαστε ότι έχουμε δουλειά που έχουμε να κάνουμε όλοι μαζί. Ο κύριος Εμμανουέλ Ιαχάν θα ξεκινήσει και μετά θα ακούσουμε όλους σας να δούμε αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες γρήγορες απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Δεν μπορείτε να απαντήσετε όλες, αλλά νομίζω ότι συναισθανόσαστε ποιε είναι οι πιο σημαντικές ερωτήσεις ο κύριος Γιάννης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να σας διαβεβαιώσω όσον αφορά την ασφάλεια των πτήσεων Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα αεροσκάφη. Είναι ένα από τα ασφαλέστερα μέση της μεταφοράς. Μπορεί να υπάρχουν σε κάποιες εταιρείες ε, ε, κάποιες καταχρήσεις εστιασμένες, αλλά η τεράστια πλειοψηφία, η τεράστια πλειοψηφία των αεροπορικών μεταφορών συμπεριλαμβανομένων και των εταιριών χαμηλού κόστου σέβονται τους κανόνες ασφαλείας και η Άσα το εξετάζει αυτό. Ε, γρήγορες απαντήσεις να δώσω. Όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείε του Περσικού κόλπου, είναι πραγματικά πρόβλημα αυτές. Έχει εκδοθεί μια έκθεση που καταδεικνύει ότι τρεις αεροπορικές εταιρείε έβαλαν ε, ερευνητές να κάνουν έρευνα και 42 δις δολάρια δόθηκαν ως κρατικές ενισχύσεις σε τρεις αεροπορικές εταιρείε, Emirates, Qatar Airways και Etihad τα τελευταία χρόνια. Για την Emirates είναι περισσότερα διότι είχαν πάρει και βοήθεια πριν ενισχύσει Για τα Emerald σήμερα είναι 59 ευρώ α380, 140 Airbus α380 έχουν παραγγείλει. σήμερα η Lufthansa έχει 15 παραγγείλει. Θα έχει 15 α380 έχει τώρα 14, έχει καμία αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, δεν έχει τα μέσα να επενδύσει ήδη ε, αυτά τα 59 δις ε, κρύβεται κάποια βοήθεια, κάποια ενίσχυση. Ε, λοιπόν, 7 με 10 φορές ο φόρος είναι πιο χαμηλός στο Αμπουντάμπι από ό,τι στην Ευρώπη. Ε, έχουμε την ίδιο ιδιοκτήτη που έχει την αεροπορική εταιρεία που έχει τις εταιρείες πετρελαίου, όχι το πετρέλαιο είναι προ, ε, ε, έχει το αεροδρόμιο ε, και έχει και τη δίκηση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Το ίδιο άτομο. Άρα καθόλου σεβαστοί κανόνες του ανταγωνισμού. Λοιπόν συνάδελφοι, λοιπόν, θα πρέπει να το καταδικήσουμε το pay to fly, αλλά δεν είναι οι περισσότερες εταιρείε που το χρησιμοποιούν αυτό και επιμένω, αν εμείς οι αεροπορικές εταιρείες Έχουμε προτεραιότητες, όπως ερωτήθηκε. Προτεραιότητα είναι ο θεμητός ανταγωνισμός. Θεμητός ανταγωνισμός τροποποιώντας τους κανονισμούς, όπως ε, και για τις εταιρείε των τρίτων χωρών. Είναι ο 648-2004 ο κανονισμός που τα διέπει αυτά. Μετά έχουμε το θέμα του σεβασμού των κοινωνικών κανόνων, πάρα πολύ σημαντικό, να καταδικάζουμε κάθε χρήση των ψευδών ανεξαρτήτων, των ψεύτικων ανεξαρτήτων και μας λένε ότι είναι αόριστο το δίκαιο κλπ. Αυτή είναι η δικαιολογία. Όχι. Αυτή η κυρία ε, Περές ε, πέρασε μια ενένεια όσον αφορά την, το μη σεβασμό ε, της απόσπασης των εργαζομένων και έχουμε συγκεκριμένο ορισμό, συγκεκριμένους ορισμούς. Από το 2002 καθορίζονται τα κριτήρια, υπάρχουν και αποφάσεις του ΔΕΚ και πρέπει να εφαρμόζουμε τους κανόνες. Νομίζω δεν εφαρμόζονται οι κανόνες. Ε, δεν είναι μόνο η Ράια. Ξέρω τον πρόεδρο της Ryanair, μου έστειλε 7 ε, επίστολες. Ε, όσον αφορά τα θέματα αυτά, γνωριζόμαστε καλά, μου ζήτησε να παραιτηθώ από τη θέση μου. Ε, υπάρχουν ποτέ δεν πήγε όταν εκδικατιζόταν οι υποθέσεις του, διότι δεν είχε δίκιο. Διότι όλες οι αποφάσεις του δικαστηρίου ε, ακολουθούσε τους κανόνες. Ένας εργο, ε, εργοδότης, ε, μία πληρωμή, μία θέση απασχόλησης. Λοιπόν, τώρα φτάνουμε στην εφαρμογή και μετά για τις τρίτε χώρες είναι το μεακό το καθεστώς που επιβάλλεται όπως είναι τα θαλασσίων μεταφορών. Αλλά ε, βρίσκουν έναν τρόπο, μας λένε ότι κανείς δεν επεξεργάζεται. Λοιπόν, βρείτε ένα τομεακό τρόπο που θα επιτρέπει τη μείωση των τελών, όπως ε, έχει ήδη γίνει στο θαλάσσιο, στις θαλάσσιες μεταφορές. Η Γαλλία χρηματοδοτεί το 74% ε, των κοινωνικών σφορών των ε, ναυτικών. Και υπάρχουν και πολλές χώρες στο 50% καλύπτουν δεν θέλουμε τέτοιου είδου κρατικέ ενισχύσει όπω τι ναυτικέ μεταφορέ, αλλά πρέπει να υπάρχουν φορολογικέ διατάξει κατάλληλε και κοινωνικέ, α πούμε, ε, τέλη του αεροδρομίου. Έχουμε ένα πακέτο για τι αεροπορικέ μεταφορέ. Στην Ευρώπη έχουμε τα πιο σημαντικά, πιο μεγάλα τέλη. Ε, συγκεκριμένα θέματα. Για την ασφάλεια των αεροδρομίων. Το ξέρετε ότι στι ΗΠΑ 60% πληρώνουν οι πολιτείε θεωρείται ότι είναι θέμα των πολιτιών και πάρα πολλές, ε, ε, σε πολλές χώρες οι χώρες πληρώνουν, όχι στην Ευρώπη, οι επιχειρήσεις που σας ψάχνουν και φροντίζουν για την ασφάλεια, που σας ψαχουλεύουν, αν, έχετε, αν κουβαλάτε κάτι παράνομο, πληρώνουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε από αυτού ε, και το Συμβούλιο δεν ήθελε να κινηθεί. Υπάρχει κάποιο κενό λοιπόν. Υπάρχει ένας τρόπος λοιπόν να βοηθήσουμε τις αεροπορικές εταιρείες να πολεμήσουν τα προβλήματα. Όσον αφορά την ε, ασφάλεια των πτήσεων, επανέρχομαι επ' αυτού. Για μας είναι σημαντικότατη η ασφάλεια των πτήσεων, αλλά η ασφάλεια των ε, πτήσεων, τι να πω, σε κάποια είδη συμβάσεων και λόγια τους ιονή ανεξαρτήτους. Σε αυτά του είδους τις συμβάσεις μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι όσον αφορά την ασφάλεια. Η ψευδής ανεξάρτητη δεν χρησιμοποιείται σαν μέθοδος από όσες αρπορικές εταιρείες, σας εξηγώ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα θέματα. Έλαβα κάποια απάντηση από την DG Moving πρόσφατα. Είχα θέσει το ερώτημα το απλό. Ε, έγινε ένα αεροπορικό δυστύχημα, Φερρυπίν. Η εταιρεία, η αεροπορική εταιρεία, έχει, έχει δύο Λέει ότι τους ασφαλίζει η εταιρεία. Ποιος είναι υπεύθυνο όμως. Η σύμβαση του Μορεάλ τι λέει. Ότι αν δεν είστε υπεύθυνο, μπορείτε να περιορίσετε την αποζημίωση που πληρώνετε στι οικογένειε στα 140 εκατομμύρια κλπ. Αν ήταν όμω ανεξάρτητοι αυτοπασχολούμενοι, θα πει η εταιρεία δεν είμαι εγώ υπεύθυνο. Δεν μου είπε ανεξάρτητο ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του. Δεν αναφέρω συγκεκριμένο ατύχημα. Αλλά θα πει δεν μου είπε τίποτα αυτοπασχολούμενο. Ο ασφαλιστή ενό ανεξαρτήτου τι θα κάνει αυτό. Θα πει περιμένετε. Η σύμβαση ε, έγινε κακή την πίστη. Πίστευα ότι ήταν ανεξάρτητος, αλλά τελικά έχει έναν μόνο εργοδότη ε, και είναι μισθωτός τελικά και όχι ε, αυτοαποσχολούμενος. Και πέρασαν 10 χρόνια, περνάνε 10 χρόνια η κατάσταση. Υπάρχουν και ένα, αλλά πρέπει να πω όμως ότι έλαβα τυχαία χθε την έκθεση. Υπάρχει επιτροπή εργασία, ομάδα εργασία που επιλαμβάνεται του θέματο και η Άζα το εξέτασε. Φοβόμασταν ότι θα πούν δεν τρέχει τίποτα και όμως θα επιληφθούν αυτού, θα δουν ποια είναι τα ρήγματα, τα κενά και υπάρχουν κράτη-μέλη των οποίων οι υπηρεσίε πολιτική αεροπορία έγραψαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπαν ότι θα πρέπει να εξεταστεί το όλο πρόβλημα. Και πιο συγκεκριμένα, υπήρχε μια ομάδα τη οποία ηγείται στη Δανία που ασχολείται με το θέμα του κοινωνικού ντάπινγκ στι αεροπορικέ μεταφορέ. Πώς ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκα περισσότερο χρόνο, την προηγούμενη φορά δεν μίλησα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι απάντησα λίγο πολύ σε όλες τις ερωτήσεις, δηλαδή έχουμε ήδη κανονισμούς, ε, το home base παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν για το home base, για την βάση για να αποφύγουμε καταχρήσεις αεροπορικές εταιρείες, όμως ε, δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Αυτά και ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Ελισαμπέτα Τσίκα. Ήθελα να μιλήσω Ιταλικά και να δώσω κάποιες απαντήσεις σε όλες τις ε, ερωτήσεις που υπευλήθησαν. Θα περιοριστώ αναφερόμενοι στο προσωπικό καμπίνας, δηλαδή στους αεροσυνοδούς ETF στις διαφάνειες έδωσε κάποιες λύσεις που θα θέλαμε να είχαμε τη δυνατότητα στο μέλλον να τις αναλύσουμε ενδελεχέστερα διότι για αυτά τα θέματα για την ώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητούμε παρά μόνο σε επίπεδο κοινωνικού διαλόγου που παρόλα αυτά είναι κάτι. Όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε περισσότερες απόψεις και με το Κοινοβούλιο και με τις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου τόσο ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις. Τώρα όσον αφορά το βασικό πρόβλημα του προσωπικού της καμπίνας, δηλαδή του outsourcing, της υπεργολαβίας του προσωπικού, πιστεύουμε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης κατάρτισης που γίνεται στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει εκεί ένα πρότυπο, στάνταρτ, συγκεκριμένο όσον αφορά αυτό. Δεν ξέρουμε πώς το προσωπικό εκπαιδεύεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το προσωπικό καμπίνα στο ευρωπαϊκό μπορεί κατά κάποιο τρόπο να αντικαθίσταται από πλήρωμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως συμβαίνει στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών όπου η πλειοψηφία του πληρώματος είναι κάτοικοι εκτός Ευρώπης, αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια των πτήσεων. Τα συνδικάτα δεν έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν την τάση όσον αφορά τις άτυπες μορφές εργασίας. Εξάλλου, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει πραγματικά μοντέλο επιβολής κυρώσεων έναντι των εταιριών που χρησιμοποιούν μοντέλα άτυπα και παράνομα εργασίας Όσα μας αφορά γνωρίζουμε η ΆΣΑ δεν έχει κάποιο μοντέλο επιβολής κυρώσεων που να μπορεί να χρησιμοποιεί να χρησιμοποιούν και εθνικοί φορείς τις εθνικές υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας και να μπορούν ε, να χρησιμοποιήσουν τις κυρώσεις ε, και να τις επιβάλλουν στις εταιρείε. Τέλος θα ήθελα να απαντήσω στον βουλευτή που έθεσε το θέμα της μητρότητας ε, των γυναικών μελών του πληρώματος είναι ένα πάρα πολύ ε, αισθητό πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε προσωπικό ε, αεροσυνοδή σε κατάσταση εγκυμοσύνης και να τις πρόχνουν σε ακραίες καταστάσεις. Δεν μιλάμε για μια απλή κοινή δουλειά, μιλάμε για μια δουλειά όπου τα άτομα κάθονται σε ένα τραπεζάκι και κάνουν μια δουλειά γραφείου. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια δουλειά που υπάρχει ανάγκη να είναι έτοιμη να κινηθεί η αεροσυνοδό σε συγκεκριμένε στιγμέ για να ανταποκριθεί και σε κατεπίγουσε ανάγκε. Αν κάτι προκύψει. Αν εκείνη τη στιγμή μια κυρία ε, ε δεν είναι σε θέση ε, να δώσει γρήγορη λύση όπω να ανοίξει μια πόρτα παραδείγματο χάρη ε, τότε η ασφάλεια της πτήσεως ε, υπονομεύεται. Ε, πιστεύω ότι να σπρώχνουμε το προσωπικό στα άκρα όπως το κάνουν κάποιες εταιρείες, δυστυχώς κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί κάποιες ευθύνες που θα πρέπει να υπομιστεί όλη η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Horn. Ευχαριστώ κύριος Χόρν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εργαζομένων στο Πιλωτήριο. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μοδοποιήσω τις ερωτήσεις. Τέθηκαν μερικέ για το ΔΟΕ, το Διεθνή Οργανισμό εργασία, το ρόλο του ε, σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η απάντηση είναι ναι ότι και ο ΔΟΕ πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο και μακάρι να έχουμε μια σύμβαση για την, για την πολιτική αεροπορία παρόμοια με αυτή που ισχύει στην αυτιλία αλλά θα είναι χρονοβόρα η διαδικασία γιατί χρειάζεται συνένεση. Έτσι λειτουργεί ο ΔΟΕ, θα χρειαστεί συνένεση μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κυβέρνηση. Και δύσκολο είναι να πιάσουμε τις κυβερνήσει κυρίε. Και τώρα ποιο ε, θα πρέπει να πρωτοστατήσει. Μα η Ευρώπη, γιατί αν δεν βάλουμε τα του οίκου, αν δεν φροντίσουμε και δεν βάλουμε μια τάξη στα του οίκου μας, πώς θα ζητήσουμε από τους εταίρους μας στην παγκόσμια κοινότητα ε, να διορθώσουν τη δική τους κατάσταση. Έχουν έχουμε ένα εναρμονισμένο νομοθετικό σύστημα και έχουμε θεσμικά όργανα που έχουν δικαίωμα δράση ε, αν έχουν και τη βούληση. Τώρα, πώς θα το καταφέρουμε. Όπως είπε κάποιος ευρωβουλευτής, έχουμε ε, υπερβολικά φιλελεύθερη γενική διεύθυνση MOVE, ιδιαίτερα για την πολιτική αεροπορία και μια λιγότερο ισχυρή γενική διεύθυνση απασχόλησης αφετέρου. Οπότε τι απομένει, θέλουμε να πρωτοστατήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπη, το προσωπικό και θέλουμε και ηγετική θέση και πίεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και να κληθούν οι αρμόδιοι να λογοδοτήσουν και να δράσουν προς σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ να αναλάβουμε τις ευθύνε μας. Τώρα, αν το πραγματοποιήσουμε, πώς θα βελτιώσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα. Φυσικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι έχει συμβεί στο πλήρωμα και στη χρήση τους. Ούτε κατά ανάγκη χρειάζεται κάτι τέτοιο πολλά, τα προβλήματα που συζητούμε. Το θέμα της έδρας βάσης, home bases, που, είναι, που βρίσκεται η πραγματική έδρα μιας αεροπορικής εταιρείας. Αυτά τα δίθεν συμβόλαια της ε, ψευτο, των ψευτοαυτοαπασχολούμενων υπάρχει ένα θέμα επιλογής, όχι πραγματικής επιλογής, δίθεν επιλογής ενός φορέα για τις απαντήσεις. Και πρέπει να πούν, εδώ είναι η έδρα, η έδρα βάσης, ε, ε, ε, εκεί είναι η η έδρα δραστηριοτήτων σα Εκεί απασχολείστε, αλλά είναι ευθέρετη ένα επιτόπου μπορεί να δούμε την πραγματικότητα, να δούμε πού απασχολείται ένα μισθωτό και να πούμε άρα αυτή είναι η έδρα βάσης. Είναι εύκολο να, πούμε, ε, να δούμε πού μια αεροπορική εταιρεία δραστηριοποιείται και να πούμε αυτή είναι η εμπορική σα έδρα και δεν σας δίνουμε αυθαίρετη επιλογή να διαλέξετε εσείς που λέτε ότι δραστηριοποιήσετε ή που λέτε ότι πηγαίνετε. Να δούμε την κατάσταση της απασχόλησης και με σαφή κριτήρια να προσδιορίσουμε αν κάποιος είναι όντως αυτοαπασχολούμενος ή ψεύτο αυτοαπασχολούμενος. Να μην αφήνουμε την αυθαίρετη επιλογή σε κάποιον υπάλληλο μια εταιρεία σε ένα γραφείο που έχει ένα όμω συμφέρον να διαλέξει την άλλη λύση. Θέλουμε σαφή κριτήρια για τα θέματα αυτά και τότε να αφήσουμε τις εταιρείε να κάνουν τι θέλουν και να αφήσουμε την κοινή λογική και τον νόμο ε, να πριτανεύσουν ε, για, το, για την εδραβάση και τους ε, ισχύοντες κανόνες. Και αν τα κάνουμε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποια στάνταρ προδιαγραφές ε, αντιμετώπισης και κανονιστικού πλαισίου χρειαζόμαστε και κάποιες διατάξεις κοινωνικής προστασίας, ε, στέγης, κοινωνικής ασφάλειας. Και αν αυτό το συνδυάσουμε με μια γνήσια αυθεντική αξιολόγηση της έδρας βάσης του home base ή της μορφής απασχόλησης, όποια και είναι η απάντηση, έχουμε προστασία και λύσεις για να, το, για να τις εφαρμόσουμε. Και ένα άλλο θέμα τώρα. Αν ε, πρέπει να διαλέξουμε τρία βασικά στοιχεία απαραίτητα για το πακέτο της πολιτικής αεροπορίας, ε, ποια είναι ε, τα πιο σημαντικά. Εγώ θα κλέψω λίγο και θα διαλέξω ένα μόνο από τα τρία. Γιατί, όπως είπαν πολλοί ευρωβουλευτές, το pay to fly και τα συμβόλαια μηδενικών ορών για για εργαζόμενους σε τόσο βασικούς τομείς ασφάλειας είναι σκανδαλώδεις μορφές. Ίσως ε, θέλετε διαβεβαιώσει, αλλά δεν πρόκειται να σας καθυσυχάσω. Είναι παραλογισμός στην αεροπορία να ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι άνω ποταμών και δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί δεν υπάρχει μία έκκληση για ολοσχερή απαγόρευση τέτοιων πρακτικών το pay to fly, του πληρώνω για να πετάξω και το συμβολέων μηδενικών ορών για απασχολούμενο σε τέτοιο κέριο κλάδο στην ασφάλεια. Μπορούμε να έχουμε μια υποχρεωτική μαθητεία ή ένα είδο ε, μαθητή για να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ τη κατάρτιση και τη ε, ε, εισαγωγή στο επάγγελμα. Αλλά όχι με αγορά πακέτο ρομπτήσεις για τέτοια κατάρτιση. Επίσης, ο κανόνας της έδρας βάσης, ένα δεύτερο θέμα ή ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούμε το καθεστώς της απασχόλησης. Να γίνει μια δίκαιη εκτίμηση του καθεστώτος απασχόλησης και όχι ένα παραπέτασμα καπνού. Επίσης το θέμα των σημειών ευκαιρίας. Πολύ σημαντικό. Ή κανόνες θεωρήσεων για το πλήρωμα που θα εργάζεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρα ε, εφαρμοστέου δικαίου να μην είναι ελεύθερη επιλογή των αεροπορικών εταιριών σε ποιο δίκαιο θα υπάγονται για να μην μπορούν να κινούνται μεταξύ διαφορετικών νομοθεσιών και να διαφεύγουν από παραθυράκια του ελέγχου και να την, να, και να επιτρέψουμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας να διαδραματίσει πιο εμφανή και ισχυρό ρόλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Τσάνβουλ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε κάποιους τομείς, να ομαδοποιήσω κάποιες από τις παρατηρήσεις μου. Συζητήθηκαν οι εντάσεις ανάμεσα στον καταναλωτή, τον εργαζόμενο, την Γενική Διεύθυνση μου, την Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση. Θα πρέπει να καταλάβουμε πώς έχει εξελιχθεί η αγορά. Όταν ξεκίνησαν Αυτές οι ε, αερογραμμές αποτελούσαν εναλλακτική λύση, πήγαιναν σε άλλα αεροδρόμια, ε, συχνά δεν είχαν βολικές ώρες, συνεπάγονταν περισσότερη μεταφορά στο έδαφος ε, του επιβάτη. Ήταν δηλαδή διαφορετική η προσφορά. Τώρα όμως όπου έχουν αναπτυχθεί, ανταγωνίζονται άμεσα τις κανονικές αεροπορικές εταιρείες ε, και πετούν από τα, βασικά, από τα μεγάλα αεροδρόμια. Σημαντικό για τους καταναλωτές είναι να έχουν πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που αγοράζουν. Εάν εσείς εδώ δεν γνωρίζετε τους όρους, ε, τότε να είστε σίγουροι ότι και ο κανονικός άνθρωπος στο δρόμο δεν θα γνωρίζει τις συνθήκες στα αεροσκάφη αυτά. Έχω φίλους που δεν είναι πολύ καλοί οδηγοί σε αυτοκίνητο. Μπορεί να μην με πειράζει να είμαι συνεπιβάτης τους ε, στην πόλη, αλλά στην εθνική δεν θα μ' άρεσε καθόλου στον αυτοκινητόδρομο. Ως καταναλωτής επιλέγω να αγοράζω τρόφιμα δίκαιου εμπορίου. Ως καταναλωτής έχω επιλογές και είναι σημαντικό να το έχουμε υποψηφτό όσον αφορά τους καταναλωτές όσον αφορά το τι μπορεί να γίνει και από το πού θα πρέπει να ξεκινήσουμε, τέθηκε το θέμα των δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην EasyJet που αναγνωρίζει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και έχει συμβάσεις ανάλογα με τη χώρα, δηλαδή οι εργαζόμενοι στην Γερμανία έχουν γερμανικά συμβόλαια σε αντίθεση με μια ε, εταιρεία όπως είναι η Ryanair. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, συχνά, ε, πρόσφατα επισήμανε τις συνθήκες εργασίας στην Ιρλανδία και ζήτησε από την Ryanair να διορθώσει την κατάσταση. Τα προβλήματα στη Δανία νομίζω δείχνουν ακριβώς τα προβλήματα αυτά. Εάν μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν επαρκή εκπροσώπηση, αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρώτο βήμα στη διαδικασία αυτή. Επίσης, υπάρχει εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την φύση των μεταφορών. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν ανάλογα προβλήματα στις οδικές μεταφορές ή στις ναυτιλιακές. Οι εργαζόμενοι έχουν μεγάλη κινητικότητα σε αυτού τους τομείς και αυτό σημαίνει ότι είναι διαφορετική τομή αυτή, είναι διαφορετικό αυτός ο τομέα ε, και ότι έχει νόημα να εξετάσουμε τους κανόνες του τομέα μεταφορών γενικά. Όπως είπαν διάφοροι υπάρχουν οργανισμοί που μπορούν να ρυθμίσουν τα θέματα αυτά και συχνά το πρόβλημα είναι η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες αυτούς. Όταν κάποιες χώρες αναλάβουν τέτοια πρωτοβουλία, οι αεροπορικές εταιρείες ε, συχνά μεταφέρουν την έδρα τους αλλού. Είναι χρήσιμο λοιπόν να υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες και ευρωπαϊκή επιβολή των κανόνων σε έναν τομέα όπως είναι οι μεταφορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκίλης και η κυρία Βάλκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να σας καθησυχάσω. Σας είπα σε κάποιον από εσά ότι μετά από την παρουσίαση που θα ακούσετε ποτέ δεν θα δείτε με τον ίδιο τρόπο τις αερομεταφορές. Θα ήθελα να τονίσω την αναφορά που έγινε στον τομέα της ναυτιλίας. Γιατί πριν την απελευθέρωση του ναυτιλιακού τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως μετά τον, πρώτο, ε, το δεύτερο ε, παγκόσμιο πόλεμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τον μεγαλύτερο στόλο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Ε, μετά την απελευθέρωση όμως ε, ο στόλος αυτός και υπάρχουν ε, πολλά θέματα ασφάλειας. Έχουμε τις ε, σημαίες ευκαιρίας Έχουμε και τα λεγόμενα πληρώματα ευκαιρίας, δηλαδή ζητάει κανείς να ζητάει τα πιο φθηνά πληρώματα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά στον κόσμο. Διότι το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκό, είναι διεθνές. Οι πρόσφατες εξελίξεις δυστυχώς μας έδειξαν την σημασία του προβλήματος. Το 44% μας είπαν ότι το καθεστώς των συναδέλφων τους ε, επηρεάζει τη διάθεσή τους να αναλάβουν μέτρα ασφαλείας. Και καθότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά είναι παγκόσμιο, ο κόσμος έχει την τάση το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και άλλοι οργανισμοί δηλαδή, τείνουν να πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μια διεθνής λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι μόνη στο θέμα αυτό. Εάν θεσπίσουμε νέους κανόνες, θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν. Κανένας δεν θα επωφεληθεί από προαιρετικούς κανόνες οι οποίοι δεν μπορούν να εφαρμοστούν κανένας ε, δεν θα υποφεληθεί από αυτό. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση την οποία ανέφερα είναι πολυτομεακή και περιλαμβάνει και όλα τα επίπεδα. Αν είναι δυνατόν το διεθνές επίπεδο, ε, τουλάχιστον το ευρωπαϊκό επίπεδο και απαιτείται ο κοινωνικός τομέας και ο τομέας των μεταφορών να συνομιλούν μεταξύ τους όπως και οι διάφορες αρμόδιες αρχές. Όπως είδαμε με τον κανόνα περί έδρας, είδαμε ότι εάν αντιγράψει κανείς μία ιδέα η οποία έχει να κάνει με την ασφάλεια και αντιγράψουμε την διάταξη αυτή σε, σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την κοινωνική ασφάλιση θα έχουμε πρόβλημα, διότι δεν είναι σαφώς ορισμένες οι διάφορες έννοιες και έτσι δεν είναι εφαρμόσιμος ο κανόνας. Το θέμα της ασφάλειας συνδέεται και με το θέμα της ευθύνης, όπως είπε ο Εμμάνουελ. Όταν έχουμε αλυσίδα εργολάβων, ποιος θα είναι αρμόδιος, σε, ποιος θα έχει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας. Ποιος θα θεωρηθεί ότι είναι ο βασικός οικονομικός φορέας. Κάτι που συνδέεται και με τον κανόνα περιέδρας. Κλείνοντας, να πω ότι πρέπει να τονιστούν τρία θέματα. Η εφαρμοστέα νομοθεσία δεν θα αντέξει στο μέλλον. Κοιτάξτε τι έγινε στον τομέα της ναυτιλίας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα και στον τομέα των αερομεταφορών. Ήδη αναζητώνται τα πληρώματα ευκαιρίε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνθρωποι δηλαδή με έδρα εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Δεύτερον, θέματα αγορά εργασία. Τα προγράμματα pay to fly θα πρέπει να απαγορευτούν. Αλλά μην ξεχνάμε, υπάρχουν επειδή υπάρχει και η αντίστοιχη αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Από ό,τι φαίνεται ο κόσμος είναι διατεθειμένος να υιοθετήσει τέτοια προγράμματα με όλα τα προβλήματα ασφαλείας που προκύπτουν. δεδομένης και τις επισφαλούς θέσης. Ε, και θα ε, επανέλθω και στην ε, βούληση των πιλότων να εφαρμόζουν μέτρα ασφαλεία όταν είναι επισφαλείς οι συνθήκες απασχόλησής τους. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το νομικό πλαίσιο, μας ενδιαφέρει και η εφαρμογή των κανόνων. Όλες οι αρμόδιες αρχές, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν πάνω στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους θερμά ε, γιατί προσπαθήσατε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, we will follow. Ε, να είστε βέβαιοι ότι θα δώσουμε συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση. Θα λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και την κατάσταση που μας παρουσιάσατε. Γιατί εδώ και χρόνια ασχολούμαστε στην Επιτροπή Απασχόληση με το τομέα των μεταφορών αλλά περισσότερο μιλούσαμε για το καποτάζ και τις οδικές μεταφορές. Και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης να εξετάσει την κατάσταση των εργασιακών συνθήκων των πιλότων, τότε και η δική μας ε, Επιτροπή άρχισε να ασχολείται και με τους άλλους κλάδους των μεταφορών. Και τα προβλήματα που έχουμε τώρα σε διάφορους τομείς των μεταφορών μας απασχολούν. Γι' αυτό και πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση. Και πάλι. Και να είναι πιο φιλόδοξη. Μάλιστα, θα οργανώσουμε και δημόσια κρόαση αργότερα, ίσως μερικοί προσκληθείτε και εκεί. Και νομίζω ότι κατέστη επιτακτική ανάγκη των αλλαγών για να αλλάξουν τα πράγματα, για να κάνουμε τη διαφορά, γιατί από όλες τις πλευρές της ε, πολιτικής αεροπορίας να βάλουμε αυτό το, μήνυμα, το μήνυμα της ανάγκης των αλλαγών. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, σας ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις που μας κάνατε και είμαι βέβαιη ότι θα ξανασυναντηθούμε. Τώρα... Σημείο 14 της ημέρης της διάταξης αποτελεσματική χρήση των πόρων και μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Θα εξετάσουμε τις 67 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο γνωμοδότησης που θα υποβάλουμε στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα δώσω τη γνώμη στην κυρία Μπέγκιν που είναι η συγγήτρια. Παρακαλώ. Grazie, signora Presidente. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις υποβληθήσεις τροπολογίες. Με τα χαράς ε, μπόρεσα να έθεσα επαφή μαζί τους και κατάφερα να λάβω υπόψη τις περισσότερες συστάσεις τους. Ελπίζω η γνωμοδότησή μας να οθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια νέα πρόταση φιλόδοξη όπως αυτή που μέχρι το τέλος του 2015 σε μια περίοδο ιστορική όπου η κρίση της απασχόλησης έχει γονατίσει πολλές χώρες, κυρίως στην Νότια Ευρώπη, η εισαγωγή ενός μοντέλου οικονομίας κυκλικής θα μπορούσε να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα. Για αυτό το σκοπό εξετίμησα τα μάλα την αναφορά στην ανάγκη να εκπαιδεύσουμε όχι μόνο τη βιομηχανία αλλά όλη την κοινωνία ούτως ώστε να καταρριφθεί το, το μοντέλο του ξέφρενου καταναλωτισμού σε πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό και αποδοτικό μοντέλο. Λοιπόν, θα ωφέλει, θα ήταν άμεσα και αυτά σε τοπικό επίπεδο, κυρίω για τι περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση και εκείνες που έχουν αισθανθεί την, τον αντίκτυπο τη αποβιομηχανοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κάτι μέλη στηρίξουν τη μετάβαση χάρη σε ευρωπαϊκέ επενδύσει, κυρίω με το ΕΦΣΥ, και να δοθούν και το Ταμείο για την Καινοτομία και θα πρέπει να προωθηθούν οι ανανεώσιμες πηχές ενέργεια και ε, να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα των αποβλήτων. Θα πρέπει να επενδύσουν ε, και ε, στους, δεν θα πρέπει να έχουμε καύση των αποβλήτων ή άλλες χωματερές. θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο την ανακύκλωση. Θα πρέπει να έχει μακρόπνο σχέδιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να μέσω της χρηματοδότησης να εγγυάται ότι οι δημόσιοι διαγωνισμοί να γίνονται σωστά και να λαμβάνονται υπόψη πτυχές κοινωνικές, περιβαλλοντικές, βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθείται η κυκλική οικονομία. Δεν θα είναι σύντομη όλη η διαδικασία, αλλά μόνο με συγκεκριμένες δράσεις μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα ήθελα να σταματήσουμε να μιλάμε και να περάσουμε στις πράξεις. Ε, έστειλε στους συναδέλφους οι γραμματεία όλες τις και περιμένω πάρα πολύ ανοιχτή και βούληση συνεργασίας ε, να ακούσω ποιε είναι οι απόψει σας και ποιε είναι οι αντιδράσει που έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την συγγήτρια, την κυρία Τιτσιάνα Μπέγκιν και τους χειόδους συγγητές και όλους τους συναδέλφους που επεξεργάστηκαν το κείμενο και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συμβούλους των πολιτικών ομάδων για τη στήριξή τους. Πολύ συχνά τους λησμονούμε και δεν τους επενούμε. Οι περισσότερες κατατεθήσεις τροπολογίες θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσε και εξυπηρετούν τη γραμμή, την πολιτική του ΕΛΚ. Θα γίνουν κάποιες προσαρμογές βέβαια για να μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνίες μεταξύ μας. Θα ήθελα όμως να σημειώσω, ενημερώνω τους συναδέρφους, ένα δισταγμό που έχω για τις παραγράφου 1 και 8 Όσον αφορά την πρώτη παράγραφο, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε συνένεση επί της ουσίας. Συμφωνούμε ότι θα ήταν κρίμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αποσύρει το νομοθετικό πακέτο που αρχικά προβλεπόταν για την κυκλική οικονομία, αλλά σημειώνουμε ότι δεσμεύτηκε να δημοσιεύσει μέχρι το τέλος του έτους μια νέα πρόταση. Θα πρέπει λοιπόν στην παράγραφο αυτή να βρούμε τα σωστά λόγια για να θετήσουμε θετική, ε, να δώσουμε θετική στάση και επικοδομητική και να μην οδηγηθούμε σε σχετισμό δυνάμεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν μα εμποδίζει να συζητήσουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και χέρια και να το ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον αφορά την παράγραφο 8, σίγουρα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μια κυκλική οικονομία, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε μια προσέγγιση πάρα πολύ περιοριστική θα πρέπει η οικονομία κυκλική να είναι ένα κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόγραμμα και να μην μεταμορφωθεί σε συμπληρωματικό κόστος για τα κράτη-μέλη που ήδη αντιμετωπίζουν ε, ανάγκες για τη μείωση του δημοσίου χρέους τους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ηλικιώτης τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, και εμεί ω ΚΟΕ πρέπει να πω είδαμε τι τροπολογίε που κατέθηκα από συναδέλφου και πρέπει να πω ότι με πολλέ από αυτέ συμφωνούμε. Ε, Κυρίω συμφωνούμε με αυτέ τι τροπολογίε οι οποίε κινούνται στην κατεύθυνση τη προστασία των εργαζομένων, όχι μόνο μέσα από συλλογικέ συμβάσει, αλλά και σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια του. Στο πακέτο των τροπολογιών υπάρχουν τέτοιε τροπολογίε τι οποίε θα στηρίξουμε, αλλά και θα τι βλέπαμε ευχαρίστω ω μέρο συμβαστικών τροπολογιών. Επίσης υπάρχουν τροπολογίες για την επανεκπαίδευση των εργαζομένων, για μέτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για δημόσιες επενδύσεις και ανάπτυξη της οικονομίας, τις οποίες θα στηρίξουμε. Δυστυχώς υπάρχει διαφωνία με όσες τροπολογίες προσπαθούν να μεταβιβάσουν τη φορολόγηση της εργασίας από τους ώμους των εργοδοτών στους ώμους των καταναλωτών. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική μια αναλογική φορολόγηση η οποία να κατανέμεται με δίκαιο τρόπο μεταξύ τη εργοδοσία του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Για αυτό το θέμα εξάλλου είχαμε καταθέσει και ανάλογη τροπολογία. Ε, Ω ΓΚΟΕ αντιλαμβανόμαστε τη σημασία τη κυκλική οικονομία για το περιβάλλον, αλλά και την προοπτική τη να δημιουργήσει θέσει εργασίε, οι οποίε όμω είναι σημαντικό να είναι ασφαλεί, αξιοπρεπεί και βιώσιμε θέσει εργασία. Και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε οικοδομητικά για συμβαστικές τροπολογίες και για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση αναφορικά με αυτήν την ε, γνωμοδέτηση. Είμαστε στη διάθεση της εισηγήτριας, την οποία ευχαριστούμε για τη δουλειά που επιτέλεσε μέχρι σήμερα και προσβλέπουμε στη μεταξύ μας εργασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Σιλικιώτη. Χρονοδιάγραμμα. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Επασχόληση Επασχόλησης χώρα στις 28 Μαΐου και στην αρμόδια καθήλια επιτροπή, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 16 με 17 Ιουνίου. Ενώ στην Ολομέλεια θα περάσει το θέμα τον Ιούλιο. Σημείο 15 της σα διάταξης, κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία για την καταπολέμηση της ανεργίας. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης, ε, της έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας που συνέταξε η κυρία Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ, στην οποία και δίνω το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντω, ε, σήμερα θα ήθελα να σα υποβάλω το σχέδιο έκθεση με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική κοινοτομία για την καταπολέμηση τη ανεργία. Πολύ σημαντικό θέμα, δεδομένου ότι η κοινωνική οικονομία είναι ένα τομέα που προσφέρει απασχόληση πάνω από 14 εκατομμύρια εργαζομένων και αντιπροσωπεύει το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δεδομένου αυτών των στοιχείων, ε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τομέα με τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης για το μέλλον. Εξού και η ανάγκη, η θεμελιώδης ανάγκη να αποφαθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά. Κατά την κατάρτιση της έκθεσής μου έλαβα υπόψη τις προτάσεις ε, πολλών οργανώσεων και συλλόγων εκπροσώπων του κλάδου και προσπάθησα να συμπεριλάβω αυτές τις ιδέες στην έκθεσή μου. Και φυσικά ε, δεσμευόμαστε από τον υποχρεωτικό αριθμό σελίδων. Αυτός μας περιορίζει και δεν μας επιτρέπει να περιλάβουμε όλα τα θέματα που θα θέλαμε, αλλά Θεωρώ ότι σε συνεργασία με τους κοιόδης και με τους υπόλοιπους ε, ευρωβουλευτές θα βελτιώσουμε το κείμενο. Μην ξεχνά την προθεσμία ε, που λήγει 21 Μαΐου 12 το μεσημέρι. Ακόμη και εγώ θα καταθέσω τραπολογίες για να βελτιώσω το κείμενο και να διορθώσω κάποια σημεία που περιλαμβάνουν σφάλματα. Καταρχήν να γίνει μια διαφοροποίηση μεταξύ των ε, επιχειρήσεων κοινωνικής ε, οικονομίας επιχειρηματικότητας από τις κλασικές επιχειρήσεις. Πολύ σημαντική αυτή η διαφορά γιατί στόχος των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας είναι κοινωνική στόχη, δηλαδή η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες, παροχή υπηρεσιών για τα μέλη τους ή δημιουργία κοινωνικού, θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου που βαίνει πέραν των στόχων των ε, συμβατικών επιχειρήσεων που στόχο έχουν κυρίως ε, την μεγιστοποίηση των κερδών τους. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η διάκριση γιατί δεν είναι το ίδιο επιχειρήσεις που έχουν κάποιες δραστηριότητες ε, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και θα πρέπει να τις στηρίξουμε και που ε, υλοποιούν και κοινωνικό στόχο και δεν έχουν μόνο εμπορικούς ε, σκοπούς. Και σε ό,τι φορά την ε, κοινωνική καινοτομία, που είναι το δεύτερο τμήμα του τίτλου της έκθεσής μου, προσπάθησα στην αιτιολογική σκέψη σίγμα τάφ την ορίσω, αλλά ως προς αυτό θα ήθελα και τη γνώμη των σχεδόν εισηγητών που να συμφωνούν με τον ορισμό που δίνω για την κοινωνική καινοτομία. Σε ό,τι τη κοινωνική οικονομία έχει πολύ σημαντικό θετικό αντικτύπο στην ε, υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής του 2020 και ιδιαίτερα στο στόχο της μείωσης της φτώχειας και της αύξησης ε, της απασχόλησης. Επίσης, επειδή δεν έχει αποκλειστικό στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους, η κοινωνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας διαθέτουν πιο μακροπρόθεσμες και μακρόπνοες στρατηγικές, ώστε τα προϊόντα τους να είναι και μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά. Οπότε η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική καινοτομία βρίσκεται ουσιαστικά στο γονιδίωμα τέτοιων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα από την ισπανική πραγματικότητα που γνωρίζω καλύτερα. Σε χώρα όπω η πατρίδα μου που έχουμε τεράστια προβλήματα υψηλής ενέργειας, όπου η κρίση υποχρέωσε ε, σε πολλές επιχειρήσεις να βάλουν λουκέτο, βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας όχι μόνο κατάφεραν να αντέξουν στην κρίση καλύτερα, αλλά από το 2008 και μετά δημιουργήθηκαν 170.000 νέες θέσεις απασχόλησης και 25.000 νέες επιχειρήσεις. Και μάλιστα στην Ισπανία σοβούζει της κρίσεις. Αυτά λοιπόν για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Και όπως αναφέρω στην έκθεση, για πολλούς και διάφορους λόγους ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε πρόσφορο έδαφος για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας για να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Οι συμβατικές επιχειρήσεις ε, έχουν ε, τα γνωστά προβλήματα και οι, κοινωνικές, οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας έχουν το επιπλέον εμπόδιο ότι δεν είναι αρκετά γνωστές και για πολλού υπάρχει αρνητική εντύπωση ότι είναι λιγότερο ανταγωνιστικέ. Θα πρέπει γι' αυτό να ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό άκθο και να βελτιώσουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων κοινωνική οικονομία στη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να προωθήσουμε τέτοιε επιχειρήσει κοινωνική οικονομία, να βελτιώσουμε τα στοιχεία που έχουμε για αυτέ και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για να δημιουργηθεί καλύτερη εντύπωση των πολιτών για τις επιχειρήσεις αυτές. Το βασικό σημείο της έκθεσης όμως αφορά τη χρηματοδότηση. Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από ότι οι παραδοσιακές συμβατικές εταιρείες. Γιατί πέραν των κονδυλίων των κοινοτικών ε, ταμείων θα πρέπει να προωθήσουμε και άλλες μορφές εναλλακτικής χρηματοδότησης, όπως είναι οι μικροχρηματοδοτήσεις ή κάποιες μορφές συλλογική χρηματοδότησης. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, να μην το ξεχνάμε, είναι, είναι σημαντικό το ταμείο αυτό και για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, κυρία Πρόεδρε, αφορά την κατάρτιση. Δηλαδή, η διαβίου κατάρτιση είναι αναφυσβήτητο ότι χρειάζεται για την καινοτομία, για την γνώση και για τη δημιουργία ειδικευμένου δυναμικού, ε, εργατικού δυναμικού. Αλλά η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να είναι η δόρατος για το μέλλον. Και αν από νωρί οι νέοι μας ε, έχουν καλή γνώμη για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία, θα είναι πολύ πιο εύκολο ε, να γίνει η κοινωνική οικονομία πιο καινοτόμα, πιο ανθεκτική και πιο ελκυστική για το μέλλον. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το πρώτο σχέδιο κειμένου. Συμμερίζομαι σε μεγάλο ποσοστό το περιεχόμενο και τις διευκρινήσεων αφορά την όλη διατύπωση. Με τα χαράς να μπορέσω να συμβάλλω και εγώ με την ομάδα μου, ο θα ξεκινήσω από ένα προβληματισμό γενικό. Κάποιε σκέψει. εκτιμώ το ότι το έγγραφο παρουσιάζει μια αξιολόγηση επίκαιρη τη σοβαρότητα τη οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και γνωρίζοντα το σοβαρό αντίκτυπο που έχει όσον αφορά τα επίπεδα τη στόχια, του κοινωνικού αποκλεισμού, τη ανεργία και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξει ρυθμό σε εθνικό επίπεδο, αλλά κυρίω σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να περάσει και πιο αποφασιστική παρέμβαση όσον αφορά τη κοινωνική οικονομία για τι επιχειρήσει και τα προγράμματα μπορούν να λειτουργήσουν με στοχευμένο τρόπο στα θέματα, στα προβλήματα τα κοινωνικά και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Η κοινωνική οικονομία πέρα από μια μέθοδο εφαρμογή ε, οικονομικών πρακτικών και επιχειρηματικότητα, πρέπει να βασίζεται επί βασικών αξιών, βιώσιμη ανάπτυξη, ένταξη κλπ. Απομακρυνόμαστε από τη λογική που επικρατεί στην κοινωνία, δηλαδή τη βελτιστοποίηση μεγιστοποίηση του κέρδους σαν μοναδικού στόχου. Αυτή είναι μια προσέγγιση που θα πρέπει να αλλάξει και πιστεύω ότι η έκθεσή μας θα πρέπει να παρουσιάζει κάποιες καλές πρακτικές του τομέα και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφέρονται οι πρακτικές και αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει στην επίτευξη του σκοπού αυτού που προανέφερα. Κεντρική σημασία είναι και η δυνατότητα των επιχειρήσεων τη κοινωνική οικονομία δημιουργούν θέσει εργασία, που σημαίνει με άλλα λόγια τη δυνατότητα μεγιστοποίηση του κοινωνικού κέρδου θα παρουσιάσω κάποιες ε, προτάσεις γι' αυτό και ελπίζω να, την, να στηρίξουν προτάσεις μου οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια Κατακλείδη κάποια διευκρίνηση επί μιας παραγράφου της 17, της παραγράφου 17 και αφορά την απέτηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει προ τι επιχειρήσει τη κοινωνική οικονομία. Πρόκειται περί ανησυχία γενική ή αναφέρεται σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων όσων σχετικές ενισχύσεις δεν δημιουργεί προβλήματα για τι επιχειρήσεις του τομέα. Εν τη αυτή περιπτώση θα ήθελα να γνωρίζω κάποιες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, Harkin. Ευχαριστώ, Marian Harkin. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη στην συγκητρία που άργησα. Διάβασα την έκθεσή σας και πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τη γενική κατεύθυνση της έκθεσης και ιδιαίτερα συμφωνώ ότι ο στόχος οποιασδήποτε κοινωνικής επιχείρησης είναι ακριβώς να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αυξήσει ε, το κέρδος της. Ε, και επίσης συμφωνώ με την θέση σας ότι με την ισχυρή τοπική τους βάση μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά οι επιχειρήσεις αυτές στην βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Κάποιες άλλες παρατηρήσεις σύντομα. Θα ήθελα κάπου στην έκθεση αυτή, αν είναι δυνατόν, να συμπεριλάβουμε την ιδέα ότι από πολιτιστικής πλευράς κάποιες ε, ιδέες περί επιχειρηματικότητας αποθαρρύνουν ε, την ανάλυση κινδύνου, αλλά συχνά οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν είναι και οι καινοτόμοι άνθρωποι, αυτοί που μπορούν να προσφέρουν νέες καινοτόμες λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε την εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας δεν πιστεύω ότι όλη η εκπαίδευση θα πρέπει να επικεντρώνεται στο θέμα αυτό, αλλά κάπου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα τέτοιο κομμάτι. Είτε συμμετέχουν σε προγράμματα οι σπουδαστές, είτε δημιουργούν μικρές δοκιμαστικές εταιρείες, δεν θα πρέπει να είναι ο στόχο τη εκπαίδευση η επιχειρηματικότητα, θα πρέπει όμως να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν και νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Επίσης, ο κόσμος όταν σκέφτεται τους επιχειρηματίες, σκέφτεται τον Bill Gates, ε, σκέφτεται τους ε, δισεκατομμυριούχους, αλλά, τους πολυδισεκατομμυριούχους, αλλά όλο και περισσότεροι επιχειρηματίε συνδυάζουν την κοινωνική και επιχειρηματική πτυχή στις επιχειρήσεις τους ε, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε και μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και στην εκπαιδευτική πτυχή διότι νομίζω ότι αυτές οι ιδέες είναι ελκυστικές για τους νέους. Μία ερώτηση για την εισηγήτρια. Στα σημεία 10 και 11 αναφέρεται στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις ε, και καλεί τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν οι κοινωνικές και κλπ. να συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις. Ερώτησή μου προς την εισηγήτρια, διότι δεν γνωρίζω πολύ καλά την οδηγία αυτή αλλά καλεί τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν κοινωνικές ρήτρε και κριτήρια τι διαδικασίε δημοσίων συμβάσεων. Ξέρω ότι το επιτρέπει αυτό η οδηγία για τι δημόσιε συμβάσει. Αλλά θέλω να ρωτήσω, τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν το κάνουν αυτό. Κάποια κράτη-μέλη βρίσκονται ε, καθοδόν. Ε, θα ήθελα την άποψή σα για το θέμα αυτό και φαντάζομαι ότι ένα από τα πράγματα που σκέφτηκα διαβάζοντας ε, το κείμενο, έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει μια γνωμοδότηση για το TTIP, αναρωτιέμαι πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, πώς θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε αυτό το μοντέλο στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας. Και τέλος, επαναλαμβάνοντας αυτό που είπε ο συνάδελφος από τους σοσιαλιστές, η συγγήτρια ζητάει ευελιξία όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, Γνωρίζω ότι έχουμε τον κανόνα αντεμήνυμης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Αναρωτιέμαι ε, αν έχει σχετικές ιδέες η συγκητρία σας. ευχαριστώ και πάλι. Είναι εξαιρετικό το κείμενο αυτό ως βάση της εργασίας μας και προσλέπω στην καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Σιλικιώτη. Κύριε Πρόεδρε, ε, καταρχήν να συγχαρώ και εγώ την συγκητρία, την κυρία Φοντάνια, για την καλή δουλειά που έχει κάνει. Ως BNGL αντιλαμβανόμαστε τη σημασία επιχειρήσεων που ονομάζονται κοινωνικές σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα πρέπει να πω ότι στη χώρα μου την Κύπρο υπάρχει ένα πολύ δυνατό κίνημα συνεργατισμού το οποίο έχει παράδοση πολλό χρόνο και το οποίο κρατά ακόμα τον ανθρώπινο του χαρακτήρα μέσα από ε, τον επιμερισμό του κοινωνικού κόστους. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να αντικαταστήσει το κοινωνικό κράτο. Το κράτο πρέπει να παραμείνει ω ο κύριος υπεύθυνο τη κοινωνική προστασία των πολιτών του, τη δημιουργία των κατάλληλων προποθέσεων για δημιουργία θέσεων εργασία και τη επανένταξη των περιθεροποιημένων ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασία. Δυστυχώ οι πολιτικέ λιτότητα που προωθούνται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τα μνημόνια και την Τρόικα, κυρίω στι χώρε του Νότου, οδηγούν σήμερα περισσότερου πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, καταστρέφοντα παράλληλα ε, νευραγικούς τομεί τη βιομηχανία των κρατών μελών, στα οποία εφαρμόζονται, διαλύοντα πολλέ φορέ κάθε ελπίδα και κοινωνική ανάπτυξη. Η ενεργή, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών μέσα από την επιχειρηματικότητα και την κοινοτομία θα μπορούσε να είναι ένα θετικό βήμα, αλλά επαναλαμβάνω Πώ την ολοκληρωμένη λύση σε αυτά τα προβλήματα μπορεί να δώσει μόνο η πολιτική δημόσιων επενδύσεων, ένα δυνατό κοινωνικό κράτο και η απαλλαγή βεβαίω από τι πολιτικέ λιτότητε. Σε ό,τι αφορά και το ερώτημα που έθεσε η εισηγήτρια για τον ορισμό τη ε, κοινωνικής καινοτομία και τη κοινωνική επιχειρηματικότητα, κατά ανάποψή μας είναι πολύ γενικό και αόριστο ε, και οι τροπολογίε που θα καταθέσουμε επί του ε, θα βασίζονται και στην ε, σημερινή μας ε, τοποθέτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you. Σας ευχαριστώ. Κάρι Μαντέλη για τους πράσινους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω την κυρία Συγήτρια για την ποιοτική της εργασία. Μια έκθεση τέτοια από το ΕΛΚ καμιά φορά μπορεί να εκπλήσει, πρέπει να το πούμε αυτό. Αισθάνομαι ότι πραγματικά κατανοήσατε το πνεύμα που δίνουμε στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και πήρατε το θέμα πραγματικά στα σοβαρά. Νομίζω όμως ότι λείπει κάπως το σφαιρικό όραμα και εξηγούμε. Για μας τους οικολόγους δεν μιλάμε κοινωνική επιχειρηματικότητα αν δεν βάλουμε και τη λέξη αλληλέγγυα. Δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Πραγματικά η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ε, ακόμα μια κάτι διακοσμητικό δίπλα στην οικονομία, την πραγματική οικονομία. Επίσης δεν είναι ειδικό τομέας που περιέχει δύο-τρεις δραστηριότητες η κοινωνική οικονομία και αλληλέγγυα οικονομία είναι εγκάρσια, μπορεί να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι κυρίως ένα μοντέλο, ένα μοντέλο που θα πρέπει να είναι ανθρώπινο, θα πρέπει να είναι συνεταιριστικό, που θα πρέπει να είναι πολύ πιο δημοκρατικό, για να το πω αλλιώς συνάδελφοι. Είναι ένα μοντέλο που προσθέτει νέες αξίες, εάν συγκρίνουμε με εκείνες τις αξίες που κυριαρχούν σήμερα στην οικονομία. Τι χαρακτηρίζει σήμερα την οικονομία. Είναι ο άγριος ανταγωνισμός, το θέμα του κοινωνικού dumping, το είδαμε αυτό στην προηγούμενη ακροασή μας, εις βάρος των γυναικών και των ανδρών, είτε είναι μισθωτοί είτε είναι καταναλωτές και δυστυχώς η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων δεν αρκεί πια. Δεν μπορεί να είναι πλέον αντίβαρο. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία θα πρέπει να είναι στην καρδιά της εκθέσεως και θα επιτρέψει να τα αλλάξουμε όλα αυτά και θα πρέπει να διαδοθεί και να εμπνέει την οικονομία μας το ταχύτερο αυτό το πνεύμα. Γιατί, διότι είναι ουσιαστικό για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, είναι η πρόκληση καταπολέμησης της ανεργίας, να φροντίσουμε ότι να είναι πιο βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, πιο σταθερές θέσεις απασχόλησης, διαρκείας και κυρίως να μην είναι, έχουμε μετακατάσταση. Η κοινωνική και αλληλέγγυα λοιπόν οικονομία είναι σημαντική πώς τι χειριζόμαστε και πώς μπορούμε να αξιολογούμε καλύτερα την οικονομία. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μας δείχνει σε ποιο βαθμό οι δείκτες μας, δεν ξέρω πώς να μεταφραστεί η λέξη που θέλω να πω στα αγγλικά, οι παρόντες δείκτες μας είναι τελικά άσχετοι θα έλεγα. Τελεί. Δεν λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα. Είναι θεροβάμονες. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους Ευρωπαίους πολίτες. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι ένας τρόπος να κινηθούμε πέρα από την απλή ανάπτυξη. Διότι ακόμα και αν η ανάπτυξη δεν έρθει, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία τελικά υλοποιείται. Αναφερθήκατε στις δυσκολίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας να βρει τη χρηματοδότηση. Πρέπει να περάσουμε πιο πέρα από αυτό. Θα πρέπει να τολμήσουμε να μιλάμε σε αυτή την Επιτροπή για το θέμα της φορολόγησης. Πολύ συχνά ανεβερόμαστε σε μια ειδική φορολόγηση για τη βοήθεια που θέλουμε να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θέτουμε βέβαια σε κάποια όρια, γιατί να μην βοηθήσουμε τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, διότι βοηθούν τους συμπολίτε μας να βρουν δουλειά και να ζήσουν καλύτερα. Το θέμα της φορολόγησης νομίζω ότι λείπει από την έκθεσή σας. Πάντως χάρη 160 ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί που εργάζονται πάνω από τον τέταρτο από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το λέω σε μια τροπολογία με αυτό για την γνωμοδότηση, για την επιχειρηματικότητα των νέων, αυτή την εβδομάδα το είπα, οι συνεταιρισμοί αξίζουν να αναγνωριστούν καλύτερα, αξίζουν πραγματικά να στηριχθούν ούτως ώστε αύριο όλο και περισσότεροι συμπολίτε μας να εργάζονται εκεί. Τέλος, μόνο 6% του ενεργού προσωπικού της Ευρώπης ζει σε αυτό το τομέα, ε, εργάζεται σε αυτό το τομέα, συγγνώμη. Χρησιμοποιείται ελάχιστα αυτός ο τομέας. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο μακριά. Γι' αυτό, και ολοκληρώνω, ολοκληρώνω, να βοηθήσουμε τους νέ, τις νέες επιχειρήσεις να παραμείνουν σταθερές. Πολλές από αυτές δεν περνάνε καν τον πρώτο χρόνο. Πρέπει να βοηθήσουμε να αντέχουν οι νέες επιχειρήσεις. Είμαι οικολόγος λοιπόν όπως σας έλεγα. Οχτώ μήνες απέχουμε από μια Διεθνή Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε ραντεβού με την ανθρωπότητα. Η Σύνοδος Κορυφής που θα γίνει στο Παρίσι και η συσχετισμός που υπάρχει μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος δεν αναφέρεται, ελάχιστα αναφέρεται στην έκθεσή σας. Η σχέση μεταξύ οικονομίας, περιβάλλοντος και πλανήτη είναι ένας μοχλός για να έχουμε μια νέα κοινωνία. Μια κοινωνία πιο αλληλέγγυα. Λοιπόν, θα πρέπει αυτοί οι στόχοι να παρουσιάζονται καλύτερα στην έκθεσή σας. Θα πρέπει ήδη λοιπόν να βασιστούμε στο σεβασμό των στόχων της κοινωνικής συνοχής, εδαφικής συνοχής, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος το ρόλο που παίζουν όλα αυτά. Λοιπόν, θα κάνω διάφορε ετοιμάσει, διάφορε τροπολογίε να σα τη δώσω για να δώσω την κατεύθυνση αυτή στην έκθεση. Σε ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω χρησιμοποίησα, έτσι. Ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ. Ο επόμενο συνάδελφο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, λέει η κυρία Μπεγκίν, όπω είπε και η κυρία ε, Φωντανιέ, η κοινωνική οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντική για περαιτέρω ανάπτυξη που θέλουμε σε περίοδο κρίσεω. Εν αναμονή εμβάθυνση κάποιων θεμάτων που αναφέρονται στην έκθεση πρωτοβουλία η συνάδελφο θα έπρεπε να τονίσει κάποιε απλέ πτυχέ. Η συγγήτρια Εν πρώτη, κάθε κράτο μέλο θα πρέπει να υποστηρίζει τι κοινωνικέ επιχειρήσει με φορολογικά κίνητρα που θα έχουν στόχο τη μείωση του κόστου εργασία και όσον αφορά την επιχειρηματικότητα την κοινωνική ε, θα, θα πρέπει να παίξουν αυτά τα στοιχεία ε, η έρευνα, επενδύσει σε έρευνα, την καινοτομία και διάδοση βελτιστών πρακτικών, που θα λάβουμε υπόψη. Υπάρχει η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική ε, ευθύνη των επιχειρήσεων διαφορετικά πράγματα. Όταν οι παραδοσιακέ επιχειρήσει εφαρμόζουν προγράμματα κοινωνικών ευθυνών τη επιχειρήση μέσω επιδίωξη κοινωνικών και περιοδικών στόχων εντό των διαφόρων προγραμμάτων των εμπορικών του και έτσι έχουν κοινωνικό αντίκτυπο όπως την μείωση της ανεργίας ίδιες επιχειρήσεις, οι παραδοσιακές ακόμα, θα έπρεπε να απολαμβάνουν από φορολογικές διευκολύνσεις που επιφυλάσσονται στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Σας ευχαριστώ. Και τώρα λόγο και πάλι στην κυρία Φοντανιά για να προσθέσει κάτι αν θέλει, μια και διατυπώθηκαν κάποιες ερωτήσεις. Μπορείτε να απαντήσετε. Έχετε την ευκαιρία τώρα. Καλώς κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ επιγραμματικά γιατί όπως διαπιστώσαμε θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για να βελτιώσουμε την έκθεση. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνεισφορά του καθενός και της κάθε πολιτικής ομάδας. Γιατί το ζήτημα αυτό για την Επιτροπή μας ε, έχει θεμελιώδη σημασία. Σε ό,τι αφορά την ε, ομιλία του σοσιαλιστού συναδέλφου συμφωνώ ότι πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Ε, για το 17 μίλησα γενικώ. Ε, και κάποιοι με του οποίου συνομίλησα μου είπαν ότι σε ορισμένε χώρες μέλη έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας που δεν ε, μπορούν να ζητήσουν ε, να καταθέσουν έτσι για ενίσχυση επειδή είχαν πολύ ε, χαμηλό αριθμό εργαζομένων. Γι' αυτό ζήτησα μεγαλύτερη ελαστικότητα. Και όταν μιλούμε για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, αν έχουν 200 εργαζομένους, αυτό είναι ένα παράδειγμα που άκουσα στο Βέλγιο. Ακόμη και με 200 εργαζομένους δεν μπορούν να ζητήσουν ενισχύσεις παρόλο που είχαν εμφανώς το χαρακτήρα των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Κυρία Χάρκιν. Περιμένω ανυπόμονα τις τροπολογίες σας και τη συνέχεια της συζήτησης. Για το TTIP και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομίζω εσείς κυρία Χάρκιν είστε πιο αρμόδια για το θέμα αυτό, είναι πιο περίπλοκο, δεν το είχα σκεφτεί είστε πλέον κατάλληλοι να το θίξετε για το πώς η συμφωνία του τύπου μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Θα ήθελα να πω στον συνάδελφο από την ΚΟΕ ότι ο ορισμός της επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας είναι περίπλοκο ζήτημα και αν θέλετε να τον αναλύσουμε περισσότερο, να το διευκρινίσουμε, γιατί όχι. Και κυρία Νταλή, Ευχαριστώ για τα ιστορικά της σχόλια. Θα ήθελα να πιστώ πω πάντως ότι η αλληλεγγύη δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της αριστεράς. Είναι κοινό μας χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, έχω παραδείγματα επιχειρήσεων κοινωνική οικονομίας της γενέτηράς μου, της Αραγώσα. Εκεί έχουμε μια συνοικία στην οποία βρίσκονται επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας γειτόνων που έχουν υποδειγματικό χαρακτήρα και δίνουν δουλειά σε πολλούς. Και μάλιστα πρόσφατα είχα συντάξει ανακοινωθέν τύπου από αυτόν τον πρόεδρο του Συλλόγου των Γειτόνων που είπε ότι από όλα τα χρόνια της δημοκρατίας ε, το πιο πρόσφορο κλίμα δημιουργούνταν επί κυβερνήσεων δεξιών του Λαϊκού Κόμματος. Οπότε η ελληνική δεν είναι ίδιον μόνο της αριστεράς, αλλά κοινό μας χαρακτηριστικό. Πάντως ε, Είμαι πεπισμένη ότι με τη συνεργασία μας θα βελτιώσουμε την έκθεση και ε, αδειμονώ για την στενότερη συνεργασία μου με τους και ηγητές. Όπως ε, προανέφερε και η κυρία Φοντανιέ, στις 21 Μαΐου το μεσημέρι λίγη προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στις 15 Ιουνίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 15 Ιουλίου. Περνάμε στο σημείο 16 τώρα. Τη μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια. Θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ζουμπέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα της φτώχειας ε, των παιδιών είναι από ίσως το μεγαλύτερο όνειδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ του 2008 και του 2012 ο αριθμός των παιδιών που ζούσαν σε οικογένειες με κίνδυνο αποκλεισμού στην Ευρώπη των 27 ε, συν Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία αυξήθηκε κατά ένα περίπου εκατομμύριο, έχοντα αυξηθεί κατά μισό εκατομμύριο μεταξύ 2011 και 2012 μόνο. Στον κίνδυνο της Ευρώ... Ε, στην Ευρώπη των 27 μεταξύ 2008 και 2012 από 26,5% αυξήθηκε σε 28%. Και το 2013, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από τη Eurostat, το 26,5 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών διέτρεχαν κίνδυνο φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού όλες οι οργανώσεις ε, χωρίς ε, καμία εξαίρεση που ασχολούνται με το θέμα αυτό και όλες οι εκθέσεις που συντάχθηκαν από ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις ε, καταλήγουν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η παιδική φτώχεια αυξήθηκε εξαιτίας κυρίως δύο παραγόντων. Έχουμε όλο και περισσότερες πολιτικές ανακατανομής του φτώχεια, δηλαδή αύξηση των, ανισο... των κοινωνικών ανισοτήτων στις διάφορες χώρες και δεύτερος παράγοντας το θέμα της πολιτικής ε, για την εργασία. Ε, με μείωση των μισθών και υποβάθμιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε πολλές χώρες, ε, ε ακολουθώντας προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικα, μειώθηκαν δραστικά οι, τα κοινωνικά επιδόματα και τα επιδόματα παιδιών. Στην πατρίδα μου την Πορτογαλία μεταξύ 2010 και 2013 Περίπου ένα εκατομμύριο παιδιά έχασαν το κοινωνικό επίδομα που ελάβαν, στα πλαίσια των οικογενειακών επιδομάτων, το επίδομα τέκνου. Και μεταξύ 10 και 2010 και 2012 περίπου 46.000 οικογένειες έχασαν το συμπληρωματικό επίδομα εισοδήματος. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες με λιγότερα παιδιά σε κατάσταση φτώχεια, δηλαδή οι χώρες, Αυστρία, Σλοβενία και Ολλανδία, είναι εκείνες που έχουν υψηλότερες κοινωνικές πολιτικές όσον αφορά την πρόσβαση στέγαση, επίδομα ανεργίας, στήριξη νηπίων, πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενώ στις χώρες που επαιδείουν λιγότερο σε αυτά τα μέτρα, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία και η Ισπανία, τα επίπεδα παιδικής φτώχειας είναι υψηλότερα. Η UNICEF αναφέρει ότι οι περικοπές του προϋπολογισμού, ιδίως στις χώρες της Μεσογείου, αύξαν την ανισότητα και συνέβαλαν στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών. Ως εκ τούτου, και αυτή είναι η γνώμη μου και αυτό λέω στην έκθεση, ότι οι πολιτικές αυτές και οι θύνοντες αυτών των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρατηγούν ή συνιστούν τον κίνδυνο παραβίασης των διεθνών υποχρεώσεων τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών ε, και του Διεθνού Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Εκπαιδευτικά ή Μορφωτικά Δικαιώματα. Οπότε, αν αυτές είναι οι αιτίες, είναι και αν ε, κάναμε σωστή διάγνωση, οφείλουμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του. Γι' αυτό και προτείνω κάποιες ε, συστάσεις. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα αναφερθώ σε ορισμένες από αυτές. Αφενός τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορέσουν να ε, προωθήσουν οικομενικά δικαιώματα για τα παιδιά και να τα σεβαστούν. Άλλωστε παρατηρούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προτείνει περικοπές στις δημόσιες δικής των αγορομελών και ε, ευελιξία στην αγορά εργασία ή ιδιωτικοποίηση των κοινοφελών υπηρεσιών. Γιατί ουσιαστικά έτσι ε, παραβιάζει την ανακοίνωση του 2013 που η ίδια υιοθέτησε για την παιδική φτώχεια. Θεωρώ επίση ότι η Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που δίνει η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου για να αυξήσουν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Παροχή Τροφίμων στου Απόρου. Και επίση ε, να θέσουν τα παιδιά ως προτεραιότητα στον προγραμματισμό και εκτέλεση των περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών συνοχής. Συστήνουμε σε όλα τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν σε όλα τα παιδιά ε, δωρεάν πρόσβαση στην παιδεία, σε παιδική παιδεία δωρεάν σε όλες τις αιτίες και να βρεθούν να βρεθού στο πλαίσιο για την παιδεία. Επίσης να, παρέχεται, να παρέχεται δωρεάν σχολικό υλικό και μεταφορά στα σχολεία. Να, να ε, εγγυθούν καθολική δημόσια δωρεάν και ποιοτική ε, υγειονομική περίθαλψη σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση, εξασφάλιση τη γυναίκα δικαιώματα σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, περίθαλψη μητρότητα κατά την προγενετική και μεταγενετική περίοδο περίθαλψη, ιδίω σε περίπτωση πρόορου του κετού, την πρόσβαση οικογενειακού γιατρού, οδοδιάτρου και ειδικού ψυχική υγεία για όλα τα παιδιά. Επίση, συνιστούμε στα κράτη-μέλη εκεί που διαπιστώνεται μεγαλύτερη ανισότητα, να ενισχυθούν τα κοινωνικά δικαιώματα και να αυξηθεί το επίπεδο ειδικών στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, αυξάνοντας την ιατρική και κοινωνική φροντίδα. Επειδή έχουμε περιορισμούς ε, ε, στο εύρος της έκθεσης, ε, δεν μπόρεσα να περιλάβω στο πρώτο μου σκαρίφημα όλες τις συστάσεις, αλλά τουλάχιστον ε, πιστεύω ότι με τις τροπολογίες θα, βελτιωθούν, θα βελτιωθεί η έκθεση, θα γεφυρωθούν τα κενά, ώστε η οριστική μας έκθεση να εντοπίζει, να κάνει διάγνωση των προβλημάτων και να προτείνει πραγματικά εναλλακτικές λύσεις και όχι τις ίδιες λύσεις ε, που ουσιαστικά ήταν η αιτία αυτού του δράματος που βιώνουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Σόιτροβα. Oui, merci, la présidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Συγήτρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας. Το θέμα αυτό της μείωσης των ανισοτήτων και κυρίως της μείωσης της στόχης των παιδιών είναι σημαντικότατο ζήτημα. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Η φτώχεια των παιδιών οδηγεί σε ανισότητες. Η μείωση των ανισοτήτων σημαίνει και μείωση της φτώχειας. Η φτώχεια των παιδιών εξαρτάται και από την κοινωνική κατάσταση της οικογένειάς τους. Από εκεί προέρχεται η φτώχεια. Η κατάσταση εξαρτάται από τα προσόντα, από την εργασία των γονέων και από τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια. Είναι και αυτό σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε την φτώχεια των παιδιών, πρέπει να επικεντρωθούμε πρώτης επί του οικογενειακού εισοδήματος. Δεύτερον, επί των δημοσίων υπηρεσιών, κυρίως επί της παιδείας. Στην έκθεση γίνεται λόγος για την αύξηση των κοινωνικών επιδομάτων και των κοινωνικών ενισχύσεων. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε περισσότερο να μιλάμε για τους γονείς που έχουν παιδιά, που εργάζονται και παρόλα αυτά βγάζουν ελάχιστα χρήματα. Ή θα πρέπει να μιλάμε για γονείς που απειλούνται από την ανεργία και δεν βρίσκουν δουλειά. Από αυτή την άποψη η απόχρωση της εκθέσεως νομίζω ότι είναι κάπως αποκλειστική ε, επικεντρώνεται επί των κρατικών ενισχύσεων και επιδομάτων. Αντιθέτως, θα προτιμούσα μια πιο πλήρη ενταξιακή προσέγγιση. Όσον αφορά την οικογένεια, βλέπω τη λύση μέσω των κοινωνικών ενισχύσεων, ίσως μικράς διαρκείας και μέτρα κοινωνικά που διευκολύνουν την κατάσταση των ε, οικογενειών, των γονέων με πολλά παιδιά και μέτρα για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των γονέων στην απασχόληση. Η κυρία Συγήτρια το ανέφερε άλλωστε. Όσον αφορά τα παιδιά, θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο επί της ποιότητας και της προσβασιμότητας στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και κυρίως πρέπει να συγκεντρωθούμε στην παιδεία, παρόλο που γνωρίζω ότι στην παράγραφο 9, 10 και 11 Μιλάμε για αυτά τα θέματα, αλλά θεωρώ ότι δεν αρκεί η διατύπωση. Θεωρώ ότι είναι εντελώς ανεπαρκή σε σχέση με τη σημασία της παιδείας, της παιδείας σαν αποφασιστικό στοιχείο για την κοινωνική κινητικότητα. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν θέλουμε να αναπαράγουμε τη φτώχεια, στις επόμενες γενιές θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί της ποιότητος της παιδείας, της εκπαιδεύσεως των παιδιών. Στην ποιότητα της κατάρτισης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποφασίζουν για το μέλλον των παιδιών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα εμπλουτίσω την έκθεση μέσω των τροπολογιών μου. Ελπίζω η έκθεσή μας να μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ευχαριστώ την κυρία Τσούμπερ για μια πολύ καλή έκθεση. Είναι σαφές το ότι ο περιορισμός όσον αφορά το μέγεθος της έκθεσης ε, την υποχρεώνει να παραλείψει σημαντικά πράγματα. Ε, ελπίζουμε να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε την έκθεση με τις τροπολογίες. Η παιδική φτώχεια είναι θέμα επώδυνο και στην Ευρώπη και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε όλα τα παιδιά. Τα παιδιά εργαζομένων αλλά και τα παιδιά ανέργων. Υπάρχουν γονείς που εργάζονται αλλά που βγάζουν τόσο λίγα που και πάλι τα παιδιά είναι φτωχά. Δεν θα πρέπει να βάλουμε σε κατηγορία τα παιδιά ανάλογα με την κατάσταση των γονιών, ε, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα παιδιά με τα ίδια κριτήρια. Στην Ευρώπη πολλές, ε, πολλοί κοινωνικοί προϋπολογισμοί έχουν βρεθεί υποπίεση, κάτι που έχει επιδεινώσει την κατάσταση πολλών παιδιών. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Τσούμπερ. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις. Ε, οι σοσιαλδημοκράτες επανειλημμένα έχουμε υποβάλει την ιδέα μιας εγγύησης για τα παιδιά. Κάτι αντίστοιχο με την εγγύηση για τους νέους να εφαρμοστούν δηλαδή ευρέως μέτρα για να καταπολεμήσουμε την παιδική φτώχεια στην Ευρώπη. Η κυρία Μπλινκεβιτσιούτη συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι χρειάζεται μία προσέγγιση που να βασίζεται στους κανόνες, ωστόσο τα αποτελέσματα της Κομισιόν του 2013 στην ανακοίνωση για τις επενδύσεις με τα παιδιά ε, επενδύσεις για τα παιδιά θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη. Οι συστάσεις είναι καλή βάση για τη δουλειά μας. Η κυρία Μπλινκεβιτσούτε θα ήθελε επίσης να τονιστεί περισσότερο το θέμα του υποσυτισμού ή της λανθασμένης διατροφής, διότι αυτό έχει σημαντικές συνέπειες για τα παιδιά. Επιπλέον η σκιώδης εισηγήτρια μας επιθυμεί να επικεντρωθούμε περισσότερο στην σημασία της εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, ε, να υπάρχει ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του και έχουμε καλές πρακτικές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν γονείς που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη από άλλους. Ε, θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Σας παρουσιάζω απλά κάποιες ιδέες της κυρίας Πλινκεβιτσιούτε, η οποία προσλέπει και στην ε, καλή συνεργασία για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε κάποιες επιπλέον ιδέες στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λιάννα Σιντάνσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια. Το θέμα αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση αυτού του θέματος. Υπάρχουν αρκετές θετικές ιδέες στην έκθεση. Μ' αρέσει η έκκληση για κοινωνικές πολιτικές στο άρθρο 8. Αποτελεί σημαντικό πρόβλημα το ότι Ε, η ταπεινή προέλευση μπορεί να οδηγήσει κάποια παιδιά σε ιδρύματα και να χάσουν τις ε, οικογένειές τους. Ε, τα παιδιά να πρέπει να πάνε σε ειδικά σχολεία επειδή προέρχονται από περιβάλλον λιγότερο ευνοϊκό. Το ότι πηγαίνουν τελικά σε ειδικό σχολείο έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη μελλοντική ζωή τους. Κάτι που λείπει από την έκθεση κατά τη γνώμη μου είναι να τονίσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και για τα παιδιά από λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα είναι τα παιδιά Ρωμά που θα ήθελα να αναφέρονται και αυτά στην έκθεση, διότι αυτή αποτελεί μία από τις βασικές μειονότητες στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν ε, την φτώχεια. Θέλουμε λοιπόν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και για τα παιδιά με αναπηρίες. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση είναι κάτι το οποίο ανέφερα ήδη κατά την πρώτη συζήτηση της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στις εξωσχολικές δραστηριότητες στα σχολεία τα παιδιά που ε, λαμβάνουν εκπαίδευση καλής ποιότητας ε, κατά τη διάρκεια των διακοπών χάνουν τις ευκαιρίες αυτές σε σύγκριση με άλλα παιδιά από οικογένειες ε, λιγότερο φτωχές. Πώς μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε τα παιδιά αυτά και κατά τη διάρκεια των διακοπών, ίσως σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε βάρος στην καλή διατροφή και στην σωστή διατροφή των παιδιών αυτών. Στη Σλοβακία πολλά παιδιά πάνε πεινασμένα στο σχολείο. Αν ε, δεν ε, λαμβάνουν ε, ένα πιάτο ζεστό φαΐ στο σχολείο, μπορεί να μην λαμβάνουν ποτέ σωστή τροφή. Ίσως λοιπόν τράπεζες τροφίμων ή άλλα μέτρα να βοηθήσουν τέτοιες οικογένειες. Σε ένα θέμα δεν συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια και ίσως να πρέπει να ρίξουμε αλλού το βάρος. Το θέμα είναι η αύξηση των επιδομάτων ανεργίας. Ωραία, θα έχουν περισσότερα χρήματα οι γονείς, αλλά τα παιδιά πρέπει να δούνε ένα θετικό πρότυπο. Θα πρέπει να δούνε τους γονείς τους να εργάζονται. Αντί λοιπόν για αύξηση του επιδόματος ανεργίας, ίσως θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον εργασίας με δημιουργία θέσεων εργασίας, ώστε οι γονείς αυτοί να μπορέσουν να βρουν δουλειά και να αποτελούν καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Αυτές είναι οι ιδέες μου αυτή τη στιγμή. Είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε μια έκθεση υψηλή ποιότητα. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κανείς από την Άλντε, ούτε από τους Πρασίνους. Από το EFTD, κυρία Πέκιν. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ τη Λαουρτζέα για την πολύ καλή έκθεση πρωτοβουλία που επεξεργάστηκε. Συμφωνούμε επί διαφόρων πτυχών που τονίστηκαν την εισηγήτρια και ιδιαίτερα μα ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Όπω υπογραμμίσαμε επανειλημμένα, ο μόνο τρόπο για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τον αποκλεισμό τον κοινωνικό είναι να δώσουμε μέτρα υποστήριξη του εισοδήματο. Μόνο εγγυόμενοι ένα ελάχιστο εισόδημα στου ε, γονείς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά εξασφαλίζοντας τη στέγη τους, την τροφή τους και την εκπαίδευσή τους. Δεν θα πρέπει να στιγματίζουμε τις Πρέπει να στιγματίσουμε μάλλον την πολιτική λιτότητα που οδήγησαν στα απελπισία και στη φτώχεια ολόκληρα, ολόκληρες ομάδες του πληθυσμού. Και τέλος πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε ε, και τις, να ε, καταπολεμήσουμε και τις νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις. Όπως η σύμβαση του αναφέρει για τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, σε όλα τα παιδιά θα πρέπει να εγγυόμεθα το δικαιώματα της εκπαίδευσης της περίθαλψης της υγείας, της στέγασης, της προστασίας, να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν, να έχουν ελεύθερο χρόνο και να μπορούν να έχουν ψυχολογικές ασχηλότητες, μία δίαιτα ισορροπημένη και ανάπτυξη εντός μιας οικογένειας. Τέτοια δικαιώματα μπορούν να προστατευτούν μόνο με, με μεγάλες επενδύσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη για το σχολείο και τη δημόσια υγεία. Ευχαριστώ ξανά την εισηγήτρια για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ετοιμάσει την έκθεση που αποτελεί αναφυσβήτητα μια έξοχη βάση εργασίας. Oh, ε, ευχαριστώ. Άρα ολοκληρώσαμε με τους ομιλητές. Εξέταση σήμερα, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ε, μέχρι 20 Μαΐου, 12 το μεσημέρι και εξέταση των τροπολογιών 15 και 16 Ιουνίου. Ενώ η ψηφοφορία θα γίνει 15 με 16 Ιουλίου στην Επιτροπή Απασχόλησης. Και φτάνουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Αλλά έχουμε, έχω κάποια προβλήματα. Πρέπει να φύγω τρέχοντας σε 10 λεπτά για να προλάβω την πτήση μου. Και είναι σημαντικό να δούμε τι θα κάνουμε με, τη, με τον προπολογισμό του 2016 και με την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Έχουμε σήμερα την πρώτη ανταλλαγή απόψεων του σχεδίου γνωμοδότησης της Τέντρε Κλούνε με θέμα την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό του 2016. Επειδή λείπει η κυρία Κλούν, θα την αντικαταστήσει η κυρία Λόπε Φοντανιά, που θα είναι όμως σύντομη. Και εγώ ερωτώ, μήπως θα μπορούσαμε να διεκπαιρεώσουμε αυτό το θέμα πολύ γρήγορα μετά την παρουσίαση της κυρίας Λόπε Φοντανιέ για να προλάβω και εγώ την πτήση μου παρά τα προβλήματα που έχω, να είμαστε λακωνικοί μετά τις παρουσιάσεις ε, και στη σχόλη έως και επιγραμματική. Ευχαριστώ. Είχε ανηλημένη υποχρέωση στην ε, Ιρλανδία κύριε Κλούν, ε, γι' αυτό και θα διαβάσω αυτά που θέλω να πει στην Επιτροπή. Παρόλο που η έκθεση για τον προπολογισμό είναι περίπλοκη, είναι σημαντικό να εκφέρουμε συνοπτική και σαφή άποψη. Επιμένουμε ιδιαίτερα στο θέμα τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων. Η ανεργία των νέων δεν είναι κάτι καινούριο στην Ευρώπη. Το 1991 είχαμε ποσοστό 21%. Έκτοτε δεν μειώθηκε ουδέποτε κάτω του 15%. Είναι αυτονόητο ότι το πρόβλημα καλύπτει ολόκληρη, αγγίζει ολόκληρη την Ευρώπη. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργία των νέων είναι 22,5% και σε μερικές χώρες μέχρι και 50%, κάτι το απαράδεκτο. Είναι σημαντικό λοιπόν να δοθεί χρηματοοικονομική ενίσχυση σε προγράμματα που επιτρέπουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με δικαιούχους ε, ε, άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Υπάρχει ανάγκη και κατάλληλη κατάρτιση και επαγγελματική ανακύκλωση σε τομεί που δεν ε, χρειάζονται εργατικό δυναμικό ή σε τομείς με μεγάλο δυναμικό όπως η πράσινη οικονομία. Πάνω από το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημιουργούν τα 2 τρίτα των, των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ δημιουργούν πάνω από το 50% της υπεραξίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τα σημαντικότερα προβλήματα για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Γι' αυτό και προτείνω αύξηση των πρακτικών και πρωτοβουλειών μικροχρηματοδότησης και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρουσιάσω τις προτεραιότητές μου. Τελεία κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που είσαστε σύντομοι. Υπάρχουν κάποιοι από τους σκιώδεις οι οποίοι θέλουν να πούν κάτι. Ορίστε. Κύριος Γκέρικε και μετά η κυρία Ζαπάλοβα. Όσον αφορά τον προπολογισμό του 2016, θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους της Ουλή και Τρεπέζιους. Ο προϋπολογισμός του 2016 αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση 26,5 δισεκατομμύρια ε, έχει ε, που δεν έχουν πληρωθεί και το ποσό αυτό θα αυξηθεί. Το χρέος αυτό είναι παράνομο και θα πρέπει να ε, πληρωθεί. Δεν επιτρέπεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκεντρώνει χρέη. Ε, στον προϋπολογισμό ζητάμε νέα προγράμματα και ε, περισσότερα χρήματα, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά η εξοικονόμηση. Μόνο στην ε, παράγραφο 3 αναφέρεται περισσότερη αποτελεσματικότητα. Ε, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται και να ε, οργανώνει νέα προγράμματα τα οποία δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει. Είναι απαραίτητο να σταματήσει αυτή η αλόγιστη δαπάνη, διότι κάθε ευρώ προέρχεται από την τσέπη των φορολογούμενων και ε, ε, αποδυναμώνει την ε, αγοραστική του δύναμη. Από πού θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μία ανάλυση των ε, αιτιών της παρούσας κρίσης και θα πρέπει να αναφερθεί εδώ η αποτυχία του ευρώ. Σας παρουσιάζω τις θέσεις της και Τρεπέζιος. Ακριβώς γι' αυτό έχουμε υψηλή ανεργία και ιδιαίτερα υψηλή ανεργία νέων. Πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συγκαλύπτουν το, ε, το πρόβλημα αυτό, προσπαθούν μάλλον να το καλύψουν χωρίς να μπορούν. Το 2014 και το 2015 δόθηκαν πολλά χρήματα για την καταπολέμηση της ε, ανεργίας των νέων και τώρα λείπουν οι πόροι αυτοί για τα επόμενα χρόνια. Η κρίση συνεχίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί εάν θέλει να συνδέσει όλα αυτά τα στήματα τόσο στενά με την ε, νομισματική ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει συνεπής εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Προγράμματα για μακροχρόνια ανέργους. Τα προγράμματα αυτά διαφέρουν πολύ εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπως ε, και τα προγράμματα κατάρτισης, μετεκπαίδευσης κλπ. Είμαστε διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν θα πρέπει να μπαίνει σε όλο και περισσότερα παιδιά τα οποία αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και που οργανώνονται μια χαρά από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη μέλη που δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά ε, σήμερα θα πρέπει να λάβουν βοήθεια για να δημιουργήσουν δικά τους συστήματα. Δεν ε, θα πρέπει όμως να βασιστούν να κάνει για αυτά τη δουλειά η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πληρωθεί από άλλα κράτη-μέλη. Δεν είναι αυτή η προσωπική μου θέση. Είναι... Σας διάβασα απλά τις θέση της κυρίας Τρεπέζιος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Τραβάλοβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρου τη συναδέρφου Ρενάτε Βέμπερ που δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα στη συζήτηση για το προϋπολογισμό του 2016. Η Συγκήτρια, ε, χαίρεται που βρίσκει τι προτεραιότητε τη ομάδα μα ε, στο σχέδιο έκθεση. Ε, ιδιαίτερα την σημασία προώθηση ε, τη επιχειρηματικότητα και των μικροβασίων επιχειρήσεων, την ανάγκη να εφαρμόσουμε αλλαγέ όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασία να ε, βοηθήσουμε την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, την ανάγκη για ε, κατάρτιση και εκπαίδευση ιδιαίτερα σε τομείς όπου δεν υπάρχει αρκετό εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, η Ρενάτε θα ήθελε να τονίσει με κάποιες τροπολογίες τις κάποιες πτυχές όπως είναι η ανάγκη όχι μόνο για σωστή ε, διαχείριση των οικονομικών, ε, αλλά να υπάρχει και αυξημένη χρηματοδότηση για το μέσο αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Η αξιοπρεπής ε, θέση εργασίας είναι ένας όρος που δεν έχει οριστεί επακριβώς. Θα θέλαμε να αντικαταστήσουμε τον όρο αυτόν με τις βιώσιμες θέσεις εργασίας. Επίσης, οι τομείς κλειδιά με σημαντικές δυνατότητες. Θα θέλαμε εδώ να προσθέσουμε και την κυκλική οικονομία στην πράσινη οικονομία ε, ε, και τις τεχνολογίες πληροφορικής ε, και επικοινωνίας, διότι μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση το 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να φροντίσουμε η να πληρωθούν οι στόχοι που αφορούν την ανεργία. Ευχαριστώ όλους και τους εισηγητές και ιδιαίτερα την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που είστε σύντομοι. Υπάρχει κανείς που οπωσδήποτε θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Να είστε σύντομος όμως. Θα προσπαθήσω να είμαι ακόμα πιο σύντομος. Καταρχάς, θεωρούμε ότι το σχέδιο εκθέσεις αποτελεί πολύ καλή βάση για τις μελλοντικές μας εργασίες. Δεύτερον, αναφέρονται σημαντικές πτυχέ που αφορούν την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσει. Δεν θα σας απαριθμίσω λόγω στενότητας χρόνου, αλλά θα σας πω τι δεν βρίσκουμε και τι θα θέλαμε να προσθεθεί. Χρειάζεται να τονίσουμε τις πηγές ε, που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους ε, του 2020 θα πρέπει να στηρίξουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και να ζητήσουμε επαρκή, επαρκή χρηματοδότηση το 2016 αναμένεται να είναι το έτος που θα έχουν ε, ξεκινήσει όλα τα προγράμματα και γενικά θα πρέπει να επιμείνουμε να έχουμε επαρκή μέτρα για να ξεπεράσουμε ε, την καθυστέρηση στις πληρωμές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για την αλληλεγγύη σας. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 13η Μαΐου το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα είναι στις 16 ε, Ιουνίου και στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού 22-23 Ιουνίου και θα γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Έτσι ολοκληρώσαμε σήμερα την ημερησία διάταξη. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου. Και ελπίζω ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε σημαντικά θέματα στις 28 Μαΐου. Σας ευχαριστώ όλους για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο.